Okay, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, then we will continue our Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα σήμερα είναι το σημείο 13 και 14 σε κοινή συζήτηση και αφορούν το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων και την σόρευση α, μεταξύ διαφόρων χωρών, συγκεκριμένα Νορβηγία και Ελβετία. Η κυρία Μπεγκίν είναι η συγγήτρια, στην οποία θα δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά τα οποία θα σας παρουσιάσω είναι δύο τεχνικά θέματα, τα οποία βέβαια είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της κοινή εμπορικής πολιτικής και πολύ ενδιαφέροντα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ουμόνων. Είναι δύο συμφωνίες, μία με την Νορβηγία και μία με την Ελβετία, που ε, τις διαπραγματευτήκαμε για τους κανόνες προέλευσης ε, στα πλαίσια του γενικευμένου σύστημα, σύστηματος προτιμήσεων. Οι κανόνες αυτοί έχουν κάνει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Τουρκία θα επιτρέπουν στις χώρες του χέρουν του γενικευμένου συστήματος να ε, εισάγουν προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, απολαμβάνοντας ε, και ε, δασμολογικές προτιμήσεις βάσει του συστήματος χάρη, υπό την προϋπόθεση ότι έχει μεταποιηθεί επαρκώς το προϊόν. Η Νορβηγία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συμφωνία και η Ελβετία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η άλλη και θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων μόνο όταν έχουν συμπεριλάβει ένα ευρωπαϊκό, ελβετικό ή νορβηγικό προϊόν στη μεταποίηση του προϊόντος τους. Αυτό έχει και αλλαγές στο σύστημα προσκόμιση αποδείξεων με την έγκριση του νέου συστήματος REX που σε κάποιες περιπτώσεις αντικαθιστά το παλιό πιστοποιητικό προέλευσης. Υπάρχει ένα κατάλογο εγγεγραμμένων παραγωγών που μπορούν να ε, παρουσιάσουν την προέλευση βάσει και της κείμενης τελωνιακής νομοθεσίας. Ξεκίνησε με ανταλλαγές επιστολών μεταξύ Νορβηγίας και Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα θα υπάρξουν αυτές οι δύο ε, συμφωνίες που απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη η έγκριση για να μπορέσουμε να έχουμε καλή ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ των χωρών και ε, μια αντίστοιχη συμφωνία με την Τουρκία δεν χρειάζεται, διότι η Τελωνιακή Ένωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Τουρκίας επιτρέπει ε, να γίνονται αυτές οι αλλαγές χωρίς να πρέπει να υπάρξει έγκριση νέα συμφωνία. Επειδή πρόκειται για τη συμφωνία δύο διεθνών συμφωνιών βάσει 200 7.4 και 208,3 της Ευρωπαϊ... Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη η συγκατάδυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Φερνάντο Περόντε Πίκνικ από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα έχω να προσθέσω στην πολύ καλή παρουσίαση της κυρίας Μπεγγέν. Να προσθέσω μόνο ότι ε, αντικαθιστούν αυτά μια συμφωνία υφιστάμενη του 2001 και πράγματι στόχο έχει να προσαρμόσει την συμφωνία στους νέους κανόνες προέλευσης ε, υπό το νέο σύστημα σε δύο τομείς. Πρώτα απ' όλα την σόρευση της προέλευσης, όπως είπαμε, μεταξύ των τριών τεσσάρων χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελβετίας, Νορβηγίας και Τουρκίας όπως και όλων των χωρών που συμμετέχουν στο γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων που άρα θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες ε, να ωφεληθούν από τις προτιμήσεις όπως ε, από ό,τι τώρα. Δεύτερον, σε σχέση με την απόδειξη της προέλευσης, θα διευκολύνει την απόδειξη προέλευσης, ε, περιλαμβάνοντας τις δηλώσεις προέλευσης από το Αρχείο Εξαγωγέων που αντικαθιστά τώρα τα πιστοποιητικά προέλευσης σε σχέση με τον χρονισμό. Ένα στοιχείο είναι ότι το νέο σύστημα αυτό υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελβετία Ελβετία και Τουρκία από πρώτης πρώτου φέτος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μόλις εγκριθούν αυτές οι προτάσεις τα πράγματα θα είναι ευκολότερα για τους εμπόρους και θα έχουμε καλύτερες συναλλαγές μεταξύ αυτών των πέντε περιοχών. Ποιος κ. δεν είναι εδώ. Τον αντικαθιστά κανείς, όχι. Χοντελίβε. Mm. Αυτή είναι η μοίρα των συντονιστών. Ο κύριος Πάμπριξ ε, απουσιάζει. Ε, δεν ξέρω, έχει γενέθλια, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μου ζήτησε όμως ε, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σύντομες. Πρώτον, ο κύριος Πάμπριξ θα ήθελε να ευχαριστήσει την κυρία Μπεγκίν για το σχέδιο έκθεσης και για την καλή του ε, συνεργασία. Ε, επί της ε, αρχής καλωσορίζει τις δύο αυτές συμφωνίες. Για να δούμε ακριβώ την επικαιροποίηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων του 2010. Θεωρεί ότι πρέπει να εγκρίνουμε και τις δύο συμφωνίες. Πρώτα απ' όλα γιατί έτσι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία και η Ελβετία να χρησιμοποιήσουν τους νέους κανόνες για την απόδειξη της προέλευσης, όπως ήδη ακούστηκε. Ένα νέο σύστημα και ελπίζουμε έτσι να αποφύγουμε και στρεβλώσεις του εμπορίου. Δεύτερον, η περίληψη της Τουρκίας στο σύστημα της όρευσης θα διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ των μερών που προαναφέραμε. Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις ε, με την Τουρκία δεν είναι στο βέλτιστο επίπεδο, γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει τουλάχιστον κάποια, υπάρχουν κάποιοι διαβλή επικοινωνίας, έστω και για τέτοια τεχνικά ζητήματα. Οπότε είμαστε υπέρ ε, των συμφωνιωθών και ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Ευχαριστώ και ο Ντάντι για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς επιτρέψτε με να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Μπεκίν για τη δουλειά που έκανε και στα δύο θέματα. Όπως υπενθύμεση σήμερα συζητάμε δύο τεχνικές συμφωνίες οι οποίες συνέφθησαν ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας και Ελβετίας για να ε, μην υπάρχει ισόρευση προϊόντων ε, από χώρες που ε, εκμεταλλεύονται το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, το GSP, δηλαδή το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προτιμησιακή μη αμοιβαία μεταχείριση για αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες. Η μεταρρύθμιση του συστήματος GSP έγινε το 2010 και προβλέπει έχουν ένα σύστημα πιστοποίηση ή πιστοποιητικών προέλευση από του ε, εγγεγραμμένου ε, ε, εξαγωγείς για να υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση. Η Ελβετία και η Νορβηγία τροποποίησαν την οδηγία του ανάλογα, την νομοθεσία του ανάλογα, συγγνώμη, για να μπορέσουν να έχουν αντίστοιχα θέματα. Όπω πολύ σωστά υπενθύμησε η συνάδελφος Μπεγκίν, η περίπτωση τη Τουρκία είναι διαφορετική, διότι η Τελωνιακή Ένωση προβλέπει τέτοια μέσα για τροποποίηση των κανόνων στην νομοθεσία, Επομένω, δεν χρειάζεται σύναψη ξεχωριστή συμφωνίας. Το νέο σύστημα προβλέπει επομένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία θα επιτρέπουν στις χώρες ε, που χαίρουν του GSP να συμπεριλαμβάνουν προϊόντα που προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα που συμμετέχει στο σύστημα, δηλαδή Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία, στην διαδικασία μεταποίησης και να εξάγονται τα τελικά προϊόντα σε κάθε μία από τις χώρες ε, που περιλαμβάνονται βάσει του συστήματος ε, GSP υπό την προπόθεση ότι έχει γίνει επαρκή μεταποίηση μεταποίηση στη χώρα προέλευση. Εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία και το γεγονός ότι έχουμε εδώ και παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να θέσω μία ερώτηση. Εχθές Είχαμε μια ενδιαφέρουσα ακρόαση εδώ στην Επιτροπή για τι μελλοντικέ εμπορικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου. Και ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν ακριβώ το θέμα των κανόνων προέλευση. Θα ήθελα να ξέρω εάν στο εγγύ μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να συνάψει αντίστοιχε συμφωνίε ε, με αυτή που συζητούμε σήμερα και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό προποθέτει. ε, ε τι, τι για τους κανόνες προέλευσης ε, και τι θα πρέπει να γίνει και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε τέτοια σημαντικά προγράμματα όπως για παράδειγμα το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων που αφορά τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ή τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την εισηγήτρια για τη δουλειά της και ελπίζω ότι το σχέδιο σύστασης θα μπορέσει να γίνει αποδεκτό με μεγάλη πλειοψηφία από την Επιτροπή και στη συνέχεια από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Thanks a lot. Uh, the other shadows are not... Ευχαριστώ. Οι άλλοι σκιώδεις ηγητέ δεν ήρθαν, δεν έχει ζητήσει κάποιον λόγο. Τον λόγο έχει λοιπόν η Κομισιόν. Έχετε κάποια σχόλια. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους βουλευτές για την πολύ ακριβή παρουσίαση των στόχων ε, και της ουσία της πρότασης Υπάρχει ένα ερώτημα όσον αφορά τις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, Βεβαίω έχουμε το θέμα των μελλοντικών σχέσεων που θα συζητηθεί σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αύριο. Ε, μετά από αυτές τις συζητήσεις θα ξέρουμε περισσότερα για το είδος της σχέσης που θα διαπραγματευτούμε. Γιατί αναλόγως με το εάν θα έχουμε μια συμφωνία ελευθεριομπορίου ή κάτι άλλο θα παίξουν διαφορετικό ρόλο οι κανόνες προέλευσης. Εν πάση περιπτώσει, εξυπακούεται ότι αν υπάρξει κάποια προτιμησιακή συμφωνία θα πρέπει να συμφωνήσουμε και προτιμησιακούς κανόνες προέλευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο και περαιτέρω συμφωνίες με άλλες ε, χώρες ε, τις οποίες δεν μπορούμε ακόμα να προδικάσουμε αλλά θα δούμε τις επόμενες ε, Εβδομάδε όσο προχωρούν οι συζητήσει. Ευχαριστώ. Ενδιαφέροντες ε, καιροί λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Και δίνω τον λόγο ξανά στην κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τη συμβολή τους. Δεν έχω και εγώ τίποτα να προσθέσω. Ας πούμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ τεχνικό και επειδή είναι και πολύ νωρίς το πρωί δεν χρειάζεται και περαιτέρω σχόλια από πλευρά συναδέλφων. Σύντομα θα πάει στην Ολομέλεια και ελπίζω σύντομα να ολοκληρώσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε και σαφείς κανόνες και για τους επιχειρηματίες μας. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίε είναι 11 ε, η ώρα στις 4 Απριλίου. Και στην επόμενη συνεδρίαση που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο θα εγκριθεί η έκθεση. Η συγγήτρια θέλει να επισπεύσουμε για την Ολομέλεια. Δηλαδή στην πρώτη ή δεύτερη Ολομέλεια του Μαΐου έχουμε προγραμματίσει να περάσει η έκθεση. Πολύ ωραία, ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το σημείο 15. Δεν βλέπω την εισηγήτρια όμως, δυστυχώς. Ελπίζω να καταφθάσει σύντομα. Αλλιώς πρέπει να αρχίσω να σας λέω αστείο. Σας λέω ανέκδοτα για να μην, μην κοιμηθείτε. Τελείωσε και το διάλειμμα. Τώρα λοιπόν σημείο 15 της Μεσαίας Διάταξης ε, είναι μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΔΕΒΕ για την διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες η περίπτωση των δασών. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις ε, για τις ε, χώρες, ε, σαν ψώμενες χώρες και την δασοκομεία και η υλοτομία εκεί, σε σχέση με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης βάσει του FLECT. Ξέρουμε υπάρχουν κάποιες χώρες που χρησιμοποιούν αυτό το πλαίσιο επιβολής της δασική νομοθεσίας τη διακυβέρνηση και το εμπόριο και ε, είχαμε μιλήσει για το φινικέλαιο και την αποψήλωση ε, των δασών στις αναψώμενες χώρες. Πολύ σημαντικό θέμα και σχετίζεται με το GSP Plus ε, και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από εκεί. Η Μαρία Αρένα είναι η εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω, η αποψήλωση, η υποβάθμιση των δασών και η παράνομη υλοτομία είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει πάρα πολλέ χώρε ανά τον κόσμο με τι οποίε έχουμε εμεί εμπειρικές σχέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή μας, στα πλαίσια αυτής της εργασίας, έχει κάθε συμφέρον να αγωνιστεί ε, κατά αυτής της αποψήλωσης, ε, διότι έχουμε απώλεια της βιοπικιλότητας ε, και υπονομεύουμε τα μέσα επιβίωσης 1,6 δισεκατομμυριών ανθρώπων, διαφθορά επίσης, βία και παραβία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι φαινόμενο που παρατηρούνται στις παραγωγικές χώρες. Η παράνομη υλοτομία και η αποψήλωση των δασών είναι εμ αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και κάποιοι από αυτούς συνδέονται με το εμπόριο. Οπότε μια εμπορική πολιτική και πολιτική επενδύσεων βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης και που εγγράφεται στα πλαίσια των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης ε, έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Από αυτή την άποψη είμαστε ο πρώτος εξαγωγέας και εισαγωγέας ε, σχετικών ε, προϊόντων και ο πρώτος εξαγωγέας ως προς τις επενδύσεις ανά τον κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ευθύνη για μια μια πιο υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση των πόρων, ε, κυρίως των δασών. για στην Επιτροπή μας ε, αυτό το δείξαμε για τα ορυκτά πολέμου, ε, στις εμπόλεμες δόνες δηλαδή. Είδαμε ποια αποτελέσματα μπορεί να έχει η πολιτική μας και σε ποιο βαθμό μπορούμε να επιβάλλουμε κάποια πρότυπα. Όμως συνιστά νομική υποχρέωση, δεν μόνο καλή πρόθεση. Ε, στο 2,15, στην 2,15 απόφαση της ε, Δικαστήριας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Σιγκαπούρης, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να σωματώσει τις αρχές της αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της βιώσιμης διαχείρισης των παγκοσμίων πόρων στην κοινή εμπορική πολιτική της, δυνάμει αυτής της απόφασης του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος σε σχέση με τις εργασίες Επιτροπής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνέπεια ω προ τι εμπορικέ πολιτικέ, πολιτικέ για τι επενδύσει, ε, καταπολέμηση τη πολυλοτομία και τη αποψήλωση ε, και βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει διάφορε δράσει ε, κατά τη παράνομη υλοτομία και τη διαχείριση των προϊόντων δασοκομεία βάσει του κανονισμού ΦΛΕΚΤΕ και στα πλαίσια των συμφωνιών εταιρική σχέση. πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε τόσο ώστε να εφαρμοστούν πλήρω αυτά τα μέτρα και να προβεί και στι απαιτούμενε αναθεωρήσει, ούτω ώστε τα μέτρα να συνάδουν πλήρω με τι διεθνεί υποχρεώσει και τι <coughs> διεθνεί και άλλε υποχρεώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, όπω ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση πρωτοβουλία το 2017 για το Φινικέλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκπονήσει ένα σχέδιο δράση για την υποβάθμιση των δασών και την αποψήλωση και την παράνομη υλοτομία, ούτω ώστε καμία αλυσίδα εφοδιασμού και καμία οικονομική συναλλαγή να μην οδηγούν σε υποβάθμιση των δασών και βλέπουμε ε, ότι <clears throat> δυστυχώ μα διαψεύδει η πραγματικότητα με αυτά που συμβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασμού του Φινίκη σήμερα λοιπόν 80% της αποψήλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο οφείλεται στην γεωργία για εξαγωγή ε, γεωργικών προϊόντων. Ε, Ω προ τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ω προ την περιβαλλοντική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο βλέπουμε ότι ε, οι πρακτικές αυτές ε, ε, είναι υπεύθυνε τουλάχιστον για το ίμιση τη αποψήλωση. Είναι λίγο ανησυχητική κατάσταση και θα πρέπει να ασχοληθούμε με, την, με αυτό το θέμα όπως και για το σόγια, το καουτσούκ, το κακάο, το βόλιο κρέα. σε χώρε με ψηλή επικλομορφία αλλά και σε χώρες με ε, ε, ε, την πρώτη ύλη που έχουν ισχυρή μεταπηκτική βιομηχανία είναι οι εταίροι μας, παραδείγματος χάρη στη Μαλαισία. Η αποψή σου οφείλεται κυρίως στο φινικέλαιο. Στην κοιλάδα του Κονγκό, παραδείγματος χάρη, πλήττεται από την αποψήλωση λόγω του καουτσούκα και για το φινικέλαιο. Το βόλιο κρέας και το, στη Βραζιλία, παραδείγματος χάρη, ε, ανάμεσα στο 2000 και 2009 το 50% ε, της ε, αποψήλωσης ήταν παράνομη υλοτομία. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε λοιπόν τη διαφθορά. Η Αργεντινή, η Βολιβία, Παραγουάη επίσης πλήττονται από αυτό το φαινόμενο τη παράνομη υλοτομία, ε, κυρίω για τη σόγια και για την εκτροφή βοήου. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσει με το Μερκοσούρ θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτέ τι προκλήσει ε, που σχετίζονται με αυτές, αυτά τα προϊόντα δοσοκομεία σε κινδύνο. Να συμπεριλάβουμε δηλαδή ένα ισχυρότερο κεφάλαιο ω προ τη βιώσιμη ανάπτυξη και εκτελεστικέ διατάξει που θα προβλέπουν και την επιβολή κυρώσεων ω ίστατο ένδικο μέσο. το ίδιο σε σχέση με την ε, η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι ο τέταρτο παγκόσμιο εισαγωγέα σε προϊόντων ξυλίας. Ε, ε, δυστυχώς η προέλευσή του ανδέχεται να είναι παράνομη υλοτομία. Ε, προς το παρόν έχουμε μόνο εθελοντικά μέτρα συνεργασία με την Ιαπωνία και αυτό οξύνει το φαινόμενο της παράνομης υλοτομία. η... Η συμφωνία σε αυτό ε, με την ε, ενίσχυση του κεφαλαίου για την βιώσιμη ανάπτυξη θα έχει σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπομειστεί τι ευθύνε τη σε σχέση ε, με αυτή την κατάσταση. Το 2013 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία μελέτη όπου βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των μεγαλύτερων καθαρού εισαγωγέ των προϊόντων αυτών που οδηγούν σε αποψήλωση 9 εκατομμυρίων εκταρίων τροπικού δάσου από το 1990 μέχρι το 2008 και αυτά λόγω της παραγωγής σόγης και καουτσούκ. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει για δυνατή προσπάθεια να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα. Η εμπορική πολιτική και η επενδυτική πολιτική είναι σημαντικό όργανα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όπως είπατε, ε, όπως και το GSP. Ε, το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στα πλαίσια ε, συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου είναι κάτι που επίσης πρέπει να ενισχυθεί και μια συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα κινδύνου είναι κάτι που θα έπρεπε να αναπτύξουμε περαιτέρω ως μέσο. Ε, θα, θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με του αρμοδίου συναδέλφου και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, γιατί είναι μέγιστε οι προκλήσει στι οποίε καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε. Ε, θα πρέπει η εμπορική πολιτική μα να γίνει ένα πραγματικό όργανο βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ένα στόχο που ανέκαθεν είχαμε εδώ πέρα στην Επιτροπή μα και ελπίζω να, να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτήν την οδό. Ε, ευχαριστούμε κυρία Ρένα. Θα ακούσουμε πρώτα του σκιώδει συζητητέ, και μετά τους, τον εισηγητή από τον από το ΕΛΚ, ο κύριος ε, Ουάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Ρούις, Ρούις με λένε, όχι Ουάς, Ρούις. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαρία Αρένα για το σχέδιο που κατέθεσε, ε, που υποβάλει, ε, την γνωμοδότηση δηλαδή που υποβάλλει προς την Επιτροπή Ανάπτυξη που είναι και η καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή, ε, θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, Ε, έχει το 4% ε, των δασών ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, το, άλλο, το υπόλοιπο 96% είναι σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτές τις χώρες ένα μεγάλο μέρος της δασοκομείας είναι παράνομη υλοτομία και έχουμε μεγάλη ευθύνη ω εισαγωγή των προϊόντων αυτή τη νοσοκομεία. Ε, Επίση, ε, πέρα από αυτό, ε, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα επί του κλίματο είναι ήδη πασιφανή και θα πρέπει να προσδιορίσουμε ένα πλαίσιο δράσης σε αυτό το τομέα και να εφαρμόσουμε ε, ένα αριθμιστικό πλαίσιο και, ένα, και μια πολιτική, μια στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της αποψήλωσης. Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη πολιτική, μια πολιτική που θα διατηρήσει, που θα προστατεύσει αυτά τα μοναδικά οικοσυστήματα. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε φιλόδοξους Στόχου ε, για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και των δασών, ε, ούτως ώστε με ισόρροπο τρόπο να ε, εκμεταλλευόμαστε τους φυσικούς πόρους. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε αυτές τις συμφωνίες για την δασική νομοθεσία διακυβέρνηση και το εμπόριο που είναι γνωστές ως συμφωνίες FLECT με το αγγλικό ακρονίμιο. Βλέπουμε ότι μπορούμε μέσω της εμπορικής πολιτικής και της επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάσουμε τις εξελίξεις σε αυτό το τομέα. διαπιστώνουμε παραδείγματο χάρη ότι υπάρχουν οι άδειε εισαγωγή. Θυμάστε ότι αρχίσαμε πριν από μία ε, δεκαετία να τις εφαρμόζουμε και έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μετά ε, ε τη, ένα χρόνο είχαμε 39.000 ε, άδειε εισαγωγή, ένα δισεκατομμύριο δηλαδή ευρώ, 25% ε, των εισαγωγών ε, προϊόντων εξηλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι έτσι μπορούμε να έχουμε ηγετικό ρόλο για την προώθηση των καλών πρακτικών, για την βιώσιμη και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων. Να ε, συνεχίσουμε την εφαρμογή, την ορθή εφαρμογή του ΦΛΕΚΤ για την ε, σωστή εκμετάλλευση των δασών, ε, να προωθήσουμε αυτές τις συμφωνίες εταιρική σχέσης με τις χώρες παραγωγούς, βασιζόμενες σε καλές πρακτικές, όπως παρατηρούμε από τις τρέχουσες συναλλαγές μας. Ε, και τώρα που συζητάμε και την στρατηγική και τα προγράμματα από το 2018 μέχρι το 2022, αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Επίσης θα πρέπει να ε, ε, εφαρμόσουμε τα κεφάλαια περί ανάπτυξης σε σχέση με όλες τις υφιστάμενες αλλά και μελλοντικέ συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Θα ήθελα ε, να ολοκληρώσω τώρα, απλώς να πω ότι θα καταθέσω κάποιες ε, τροπολογίες ε, για το σχέδιο της κυρίας Αρένα. Πάντως, της ευχαριστώ όλους ιδιαίτερως για το περιεχόμενο της εκθέσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Γουίς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την εισηγητρία για τη δουλειά που έκανε και την συνεισφορά της. Σ' ονόματος της Άλτα... θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Επηρεάζει βεβαίως και την κλιματική αλλαγή. Είναι αποφασιστικό να υπάρχει βιώσιμη δασοκομεία και πρέπει να το τονίσουμε αυτό και στις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις. Βεβαίω οι εφοδιαστικές αλυσίδες ε, έχουν μεγάλη σημασία, όπως έχει σημασία και η εφαρμογή των διατάξεων. Εφαρμόσιμες λοιπόν διατάξεις ε, για να είμαστε σίγουροι ότι θα ισχύσουν. Οπότε το νόημα δεν έχει να βάλουμε εδώ πέρα ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και να έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι έφικτα, αλλιώς απλούστατα θα αγνοηθούν. όπως είπα λοιπόν, να είναι εφαρμόσιμα. Αναμένουμε λοιπόν την συνεργασία στο σημαντικό αυτό θέμα και Νομίζω τελικά θα καταφέρουμε κάτι καλό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τους πράσινους και την Κούε δεν είναι κανείς. Α, ο Χέλμουτ. Ναι, αντικαθίστω την κυρία Σάντσες που κολλείεται. Μου ζήτησε να μεταφέρω κάποια λόγια. Η Λούλα Σάντσες Ευχαριστή λοιπόν την εισηγήτρια για την ε, δουλειά που έχει κάνει. Θεωρεί ότι πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα προωθήσουμε μια πιο βιώσιμη διαχείριση των δασών στις αναψώμενες ε, χώρες. Έχουμε 8,8 εκατομμύρια εκταρίων ε, κάθε χρόνο που χάνονται και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ένα σχέδιο δράσης το οποίο οδήγησε στην αύξηση των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς ε, έχουμε την ε, εκμετάλλευση των δασών ε, και την αποδάσωση και ανησυχώ ιδιαιτέρως, λέει η κυρία Λούλα Σάντσες, πως πάρα πολύ συχνά οι διαβουλεύσει με την κοινωνία των πολιτών, τους ηθαγενείς και τους εργαζόμενους συχνά είναι ανεπαρκείς. Έτσι μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να τονίσουμε την σημασία αυτών των διαβουλεύσεων με επαρκή ενημέρωση και ελευθερία απόφασης τέλος η ομάδα μας ε, θα καταθέσει κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Κάποιες πτυχές δηλαδή της έκθεσης που θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάνε προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Και βέβαια αναμένουμε τη συνεργασία με την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα η Χάιντι Χάουταλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερο. για το ότι οι τρεις επιτροπές ε, και η Διεθνούς Εμπορίου και η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, και η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, να συντάξουν αυτή την έκθεση με βάση το άρθρο 54 Υπάρχει λοιπόν μια καλή κατανομή εργασίας. Υπάρχει όμως περιθώριο για την Επιτροπή Διεθνού Υπορείου να οφήσει την έκθεση αυτή. Μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που είναι νομίζω επικαιρή. Γιατί θα δημοσφάνει μόλις τώρα η Κομισιόν ε, και από το Κοινοβούλιο να συντάξει ένα σχέδιο δράσης για την αποδάσωση και την Παρασκευή που μας πέρασε η Κομισιόν ε, δημοσίευσε μια μελέτη που έχει στόχο ακριβώς ε, να συντάξει το σχέδιο δράσης και βλέπουμε εδώ πέρα από τη μελέτη αυτή πως υπάρχουν πολλές επιλογές για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει την αποδάσωση και ενδιαφέρον είναι πως ε, πολλές από αυτές τις ε, συστάσεις ε, εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Γιατί αναφέρεται εδώ πέρα το ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ιδέουσα επιμέλεια. Κάτι το οποίο ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο είπε η Μαρία Αρένα, ότι πρέπει να προτείνουμε Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να μπορέσουμε να δούμε και τις συμφωνίες αυτές τις εθελοντικές και θεωρώ ότι θα πρέπει και η Επιτροπή μας να εκφράσει την άποψη της. Γνωρίζω πως από τις 16 συμφωνίες οι διοικητικοί πόροι στις, στην Κομισιόν και στις αντιπροσωπείες δεν επαρκούν για να δουν εάν εφαρμόζονται. Το ένα είναι αυτό. Θα έλεγα ότι το θέμα των βιώσιμων ε, εφοδιαστικών αλυσίδων σχετίζεται με το ότι τα δάση παραγούν ε, διάφορες αξίες και προσθέτουν αξία και μπορεί έτσι να βγάλουν το βιός τους ε, πολλοί άνθρωποι και αυτόχθονες ε, πληθυσμοί. Εάν ε, μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε λοιπόν μια τέτοια βιώσιμη διαχείριση για να έχουν και δουλειές οι άνθρωποι που ζουν κοντά στο δάσος νομίζω ότι έτσι θα προωθήσουμε τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης. Βεβαίω πρέπει να δούμε και τις ε, μεγάλες φυτίες ε, και τον ρόλο που παίζουν ε, στα δάση. με την αποδάσωση αλλά και το πως οι τοπικοί πληθυσμοί μπορούν να ενθαρρυνθούν να προστατεύσουν το δάσος έχοντας και οικονομικά ωφέλη. Μεγάλη σημασία λοιπόν εδώ πέρα η εφοδιαστική αλυσίδα. Πολλά δάση κινδυνεύουν, δεν έχουν την σωστή διαχείριση. Αυτό σχετίζεται και με τα συστήματα διακυβέρνησης. Αν ενισχύσουμε λοιπόν τις σχετικές πτυχές, ειδικά όπως πρότεινε η Μαρία Αρένα, στα σχετικά κεφάλαια, θα είναι κάτι το εξαιρετικό. Και τώρα που είδαμε όλες αυτές τις αντιδράσεις από τις χώρες που παράγουν φίνη και ελαιό αντιδράσεις απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους εμπορικούς μας εταίρους για να φροντίσουμε οι δασοκομικές πρακτικές τους να μην επιταχύνουν την αποδάσωση και την αποψήλωση των δασών. Μπορούμε πράγματι να ε, ενισχύσουμε ακριβώ και το βιός των ανθρώπων που ζουν από το δάσος. Ε, δεν είναι, αυτά τα πράγματα δεν είναι αντιφατικά. Θα έλεγα ότι πάνε χέρι με χέρι. Θα έχουμε λοιπόν μια σημαντική συνεισφορά του Κοινοβουλίου Ε, για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το σχέδιο δράσης ε, για την αποδάσωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, Έμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, στη Μαρία Ρενά, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά είναι εξαιρετική η γνωμοδότηση και θα ήθελα να εστιάσω σε μια πτυχή που ανέφερε συνάδελφος από τους φιλελευθέρους για τον έλεγχο της εφαρμογής και υλοποίησης των μέτρων και κυρίως της πιστοποίησης ξυλίας ε, από δάση ε, για νόμιμη υλοτομία. Διότι από κάποιες πληροφορίες ε, στις οποίες είχα πρόσβαση, θεωρώ ότι δεν γίνεται παρκής έλεγχος ε, για τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται τα πιστοποιητικά ε, σε κάποιες επιχειρήσεις και τελικά φτάνει στις αγορές μας ξυλία από δάση που έχει μεν σωστή πιστοποίηση αλλά δεν ανταποκρίνεται ε, σε νόμιμη υλοτομία. Επομένως θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο γεγονός αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γνωστή ε, εταίρος μας, η Μαντλέν. Ε, τι πιστεύετε ότι σας βοηθάμε λίγο με αυτά τις κατευθυντήριες γραμμές ε, που δίνουμε. Ε, καλά κάνατε και αποφύγατε κι εσείς το επίθετό μου και εγώ το ίδιο κάνω. Ε, ευχαριστώ. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την παρουσίαση από την κυρία Αρένα και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων για τις σχέσεις ανάμεσα στη, στα δάση και το εμπόριο. Ε, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων ε, με σχετίζεται με πολύ ενδιαφέρον τρόπο με το εμπόριο όταν μιλάμε για τα δάση. Ε, μιλάμε για ε, καθαρό εξαγωγέα, προ, εισαγωγέα προϊόντων ε, Έχουμε αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες όπως το ΦΛΕΚΤΕ για την ε, βιώσιμη διαχείριση των προϊόντων εξηλίας, ε, για την ε, παράνομη υλοτομία και σχετικέ σχετικές εμπορικές σχέσεις. Έχουμε πρακτικές που έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια και μέσα στις εμπορικές συμφωνίες με τα κεφάλαια βιώσιμης διαχείρισης και συγκεκριμένα με το πλαίσιο ΦΛΕΚΤΕ και τα κεφάλαια TST. Εύχομαι. Τώρα, σε σχέση με τον κίνδυνο να εφαρμόσετε τα μέτρα για ε, κάποια προϊόντα και όχι άλλα και να μην συμφωνούμαστε με τις διεθνείς ε, υποχρεώσεις, ε, προσπαθούμε να κάνουμε τακτικές αναθεωρήσεις. Υπάρχει το θέμα της δέουσας επιμελητίας, διότι μιλάμε και για πρώτα όπως τα κλωστεφαντουργικά. Το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε, έδωσε την έγκρισή του για μια οδηγία για την παραγωγή οικονομικών πληροφοριών από πλευρά των επιχειρήσεων, παραδείγματο χάρη ε, οι επιχειρήσεις ε, πρέπει να δίνουν τώρα στοιχεία για τη βιωσιμότητα της ε, πολιτικής τους μέσα στις οικονομικές τους εκθέσεις. Θα δούμε τώρα με αυτή τη διαφάνεια αν τελικά θα υλοποιήσουμε τον στόχο που έχουμε θέσει. Η διαφανής και η υπεύθυνη βιώσιμη διαχείριση των ε, δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες και η σχέση της με το εμπόριο, ε, τι να σας πω, ελπίζω ε, η Επιτροπή να αναγνωρίσει τη χρησιμότητα των εργαλείων που έχουμε ήδη ε, στο πλωστάσιό μας, καθώς να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε το μίσο όπου ενδεχομένως μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν επίσης σε πρόσφατες ε, μελέτες, οι ε, ανεξάρτητες μελέτες ε, που δημοσιεύθηκαν για τη μορισιμότητα του εμπορίου του φινικελαίου και για τα διάφορα προϊόντα που έχουν εκπονηθεί από εμπειρογνώμονες μετά από δικό μας έτοιμο θα αξιολογήσουμε το περιεχόμενό τους και θα κρίνουμε αν θα πρέπει να ληφθεί μελλοντικά δράση για, κατά της παράνομες υλοτομίας και της αποψήλωσης. Ε, πολλά σημεία είναι ιδιαίτερα τεχνικά, οπότε με χαρά να συνεργαστούμε διμερώς μετά την συνεδρία. Σε ευχαριστούμε. Thanks a lot. Uh, on the issue. Ευχαριστούμε για το θέμα FLECT. Μου δίνετε και κάποια ε, στοιχεία. Ε, πόσες χώρες, ας πούμε, χρησιμοποιούν ε, το FLECT. Και γενικά ποιες εμπειρίες έχουμε μέχρι στιγμής από την εφαρμογή του FLECT. Εγώ είμαι από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπόριο και είναι κοινό το θέμα. Εγώ τα είπα τα εμπορικά ζητήματα και θα δώσω το λόγο στην άλλη από την ΤΕΦΚΟ. Μάριο. Μαρία. Μαρία Πάρτα από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΤΕΦΚΟ. Καλημέρα. Αν κατάλαβα καλά τι μας ρωτάτε, ε, πόσες χώρες ε, ε, εξάγουν ε, ε, δαλία, εξηλία συγγνώμη, με άδεια φλέκτε, μόνο μία, η Ινδονησία. 40.000 άδειε μέσα σε ένα χρόνο. Είπαμε ένα δις δολάρια ήταν η αξία αυτών των αδειών. Η Γκάνα αναμένεται να προσχωρήσει σε αυτή την ομάδα πιστοποιητικών φλέκτ. Όχι φέτος, του, του χρόνου περιμένουμε τέτοιε εξαγωγικέ άδειε για την Κάνα. μπορείτε λίγο να μας μιλήσετε για τα προβλήματα. Γιατί, γιατί καθυστερούμε τόσο πολύ με αυτή τη διαδικασία. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και μπορεί να χρειαστώ πολύ χρόνο για να σας εξηγήσω ακριβώς τις προκλήσεις. Η Γκάνα ε, ήταν η πρώτη χώρα που υπέγραψε το 2009 μια VPM μια θελοντική τέτοια συμφωνία. Η Ινδονησία πολύ αργότερα. Στο μεταξύ έχουμε και άλλες 9 χώρες ε, που εφαρμόζουν τις VPAs ε, και 6 ακόμη με τις οποίες διαπραγματευόμαστε ε, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Νοτιοανατολική Ασία είναι αυτές οι χώρες. Το FLEC και VPAs, οι δημοτικές συμφωνίες δεν σχετίζονται μόνο με το εμπόριο αλλά και με τη διακυβέρνηση. Δύσκολα, δύσκολες οι συνθήκες διότι θέλουμε να αναβαθμίσουμε την ε, διακυβέρνηση, τη διαφάνεια, την ε, συμμετοχή, τη λογοδοσία, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο, στο φλέκτ και δεν τα καταφέρνουμε πάντοτε ε, όπως θα θέλαμε. Παραδείγματος χάρη για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Η ξυλία αυτή τη στιγμή συνδέεται με τις ε, σειράξεις. Αναβιώσαμε τη διαδικασία φλέκτ για να Υπάρχει ένας ε, χώρος ε, για να γίνει ο διάλογος για την ε, διακυβέρνηση και τη διαφάνεια, αλλά θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα συζητάμε για την ξυλία στο Κονγκό. Στη Λιβυρία μετά, τη... μετά σειραξιακή χώρα, εξαιρετικά εύθραυστη, πολύ δύσκολο πρόθεσμα να έχει κάποιος αυτά αποτελέσματα από τέτοιους διαλόγους. Ε, τώρα επεξεργαζόμαστε ένα ε, σχέδιο εργασίας για τις νέες θελοντικές συμφωνίες που ελπίζουμε να ε, προτείνουμε στο Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του τρέχοντος. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, θέλω να επιστρέψω στο θέμα του Φινικελαίου. Μπορείτε να σχολιάσετε αυτή την αντίδραση που τη σκληρή αντίδραση της Μαλαισίας και της Ινδονησίας. Μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Χάιντι Χάουτελα. Δεν είναι εύκολο, είναι εξαιρετικά περίπλοκο το ζήτημα της αποψήλωσης. Γι' αυτό κάναμε δύο μελέτες αντικτύπου που έχουν δημοσιευθεί και θα μας δώσουν στοιχεία για να, να λάβουμε τη βέλτιστη δυνατή δράση επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ήταν ε, πολύ ισχυρές ε, ε, αντιδράσεις ε, γιατί από πλευράς Μαλαισίας και Ινδονησίας και πρέπει να δούμε ε, πώς θα περάσουμε από την παράνομη στην νόμιμη υλοτομία με το σχέδιο δράση. Είναι ιδιαίτερα καθόδες το πολιτικό αυτό ζήτημα και όχι μόνο σε σχέση με αυτές τις δύο χώρες αλλά και από την άλλη πλευρά με τη Βραζιλία. Ναι και με το Περού ήταν καυτό το ζήτημα Σόλτ και Χάουτελ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δύο επιπλέον εξηγήσει. Ε, αυτό βέβαια μας οδηγεί και ακριβώς ε, στο μέχρι ποιο σημείο ε, το σύνθετο και περίπλοκο θέμα της διακυβέρνησης που μόλις μας περιγράψετε συμπεριλαμβάνεται στις ε, διαπραγματεύσεις ε, ελευθέρων συναλλαγών ε, για το φινικέλαιο, τι κάνετε με τη Συμφωνία Μερκοσούρ και που βλέπετε και την ευθύνη να το συμπεριλάβουμε όλο αυτό στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Δεν αρκεί το γεγονός ότι υπάρχει σχετικό κεφάλαιο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλα αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα και προκλήσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για χώρες ε, με τις οποίες δεν έχουμε διευρυμένες εμπορικές ε, σχέσεις. Για παράδειγμα, η Ρωσική Ομοσπονδία έχει σοβαρά θέματα δασών ε, και δεν έχουμε πάει πουθενά μαζί τους. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και τις συμφωνίες FLEGD για να στρέψουμε και το βλέμμα μας προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Χάουταλα, που εξήγησε τα θέματα αυτά. Έχω κάποιες περαιτέρω ερωτήσεις. Ε, πολύ σωστά αναφέρεται ότι υπάρχουν εργαλεία και ότι συζητάμε αυτά τα εργαλεία και υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Ε, το δικαίωμα γιατί που υπάρχουν τώρα, τα δικαιώματα που υπάρχουν τώρα, η εντύπωσή μου είναι ότι τα θέματα διακυβέρνησης και αυτό που ε, αποκαλούμε έμεσες συνέπειες χρήσης γης ε, δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη σε αυτά τα μέσα, για παράδειγμα στις ε, θελοντικές συμφωνίες εταιρική σχέσης. Είναι σωστό αυτό, μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το τομέα. Και δεύτερη ερώτηση, ε, θεωρείτε ότι αυτές οι εθελοντικές συμφωνίες εταιρικές σχέσεις βοηθούν να έχουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας στον τομέα των δασών. Uh, Ποιο θέλει να απαντήσει, παρακαλώ. Νομίζω ε, θα απαντήσουμε εδώ ντουέτο. Η πρώτη ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί σε δύο λεπτά ε, το κατά πόσο η διακυβέρνηση περιλαμβάνεται στις ε, διαπραγματεύσεις στην εξελίξη. Είναι σαφές ότι Έχουμε να κάνουμε εδώ με διαχείριση γεών και είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. Οι συζητήσει είναι εν εξελίξη, κυρίω με τι δύο χώρε με τι οποίε διαπραγματευόμαστε για το φινικέλαιο. Δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμα την απάντηση και κάποιε από τι αντιδράσει στι οποίε αναφερθήκατε, ιδίω στην Ινδονησία και στη Μαλαισία, αντανακλούν ακριβώ τι προκλήσει στο εμπόριο και εμπορικού όρου ε, που δεν μπορούμε να ε, διακρίνουμε για παραπροϊόντα. Εάν λάβουμε υπόψη μας το φινικέλαιο, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελεί διάκριση γιατί δεν θα λάβουμε υπόψη κάποια άλλα προϊόντα. Είναι σαφές ότι με την Ινδονησία θα χρειαστούμε μία λύση με το φινικέλαιο και αυτό το οποίο πρέπει να δούμε σε εσωτερικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τι ισχύει για την ε, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Η Μαρία θα απαντήσει το θέμα για τη διακυβέρνηση και τις ε, συμφωνίες ε, τερικής σχέσης τις εθελοντικές. Δύο θέματα για αυτές τις συμφωνίες. Η διακυβέρνηση είναι ο πυλώνα της δράσης FLEGD, είναι πολιτικά σημαντικό πυλώνας των εθελοντικών συμφωνιών και είναι η σημαντική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για να δίνονται οι άδειε διαφάνεια, λογοδοσία, συμμετοχή, καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, σημαντικά στοιχεία λοιπόν τα οποία μας απασχολούν με τις χώρες εταίρους προκειμένου να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και να καταλήξουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Βέβαια ούτε το FLEGD ούτε οι συμφωνίες ε, αυτές οι εθελοντικές ε, αποτελούν πανάκια για τα πάντα. Η ε, βιώσιμη διαχείριση των δασών είναι η μακροπρόθεσμη στόχη και προσπαθούμε μέσω του FLEGD, μέσω των συμφωνιών αυτών να δημιουργήσουμε το κατάλληλο χώρο για διάλογο για να γίνει ο διάλογος σε εθνικό επίπεδο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και βλέπουμε ήδη ότι υπάρχουν αρκετά σημεία πρόοδου για παράδειγμα, στι τρέχουσε διαπραγματεύσεις με την Ονδούρα και την ε, ε Φαίνεται ότι έχουμε καταλήξει συμφωνία και με τις δύο χώρες για να υπάρχει μια αρχή μη διάκριση στις εθελοντικέ συμφωνίε τερικέ σχέσει όσον αφορά τους ε, διαφόρους ε, ενδιαφερομένους και τα αγαθά που παράγουν οι αυτόχθονε πληθυσμοί καθώς επίσης και στην Γουιάννα που ε, η χρήση γεών ε, από τους αυτόχθονες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ε, συμφωνήσαμε να συμπεριλάβουμε και ένα μηχανισμό που θα επιτρέψει και στην κυβέρνηση και στους αυτόχθονες πληθυσμούς να συζητήσουν τα θέματα και άλλους ενδιαφερομένους βεβαίως να συζητήσουν τα θέματα και να επιλύσουν το ζήτημα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτές τις εθελοντικές συμφωνίες για να δημιουργήσουμε το περιθώριο για να γίνουν αυτές οι συζητήσει και ενδεχομένως να επιληθούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά οι εθελοντικέ συμφωνίε εταιρικέ σχέσεις δεν είναι το μέσο για να επιλύσουμε τα πάντα. Ευχαριστώ και για να ολοκληρώσουμε η συγγήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι ήδη στα πλαίσια της σημερινής συζήτησης διαπιστώνουμε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα και ε, το γεγονό ότι πρέπει να το προσεγγίσουμε συνολικά το θέμα της αποψήλωση. Όπως ε, είπα προηγουμένως και στην παρέμβασή μου, η αποψήλωση δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο εμπόριο ξυλία. εξαρτάται από το εμπόριο ξυλία και φυσικά και από την παράνομη υλοτιμία, αλλά όσον αφορά την νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, Πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση της νομοθεσίας, εφαρμογή του κανονισμού και να δούμε και τι συνοδευτικά μέτρα ε, έχουν εφαρμοστεί και να αξιολογηθούν και στις συμφωνίες FLECT ε, και στις ενθελοντικές συμφωνίες. Αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά την παράνομη αλυσίδα εξαγωγή και μεταπλήρωση ξύλια. Άλλωστε με εκπλήσει το γεγονό ότι η Γενική Διεύθυνση Ταξούντ δεν είναι παρούσα εδώ. Γιατί ένα από του λόγου για του οποίου υπάρχει και αυτό το θέμα τη παράνομη αλυσίδα ε, ξυλία είναι γιατί στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρουμε να ελέγξουμε σωστά αυτό που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες φορές εμένα με εκπλήσει αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι η νομοθεσία για τη διαμάντη είναι δύσκολα γιατί το κρύβει κάποιος, εύκολα το διαβάνει. Αλλά ε, κορμούς ξύλου, τεράστια <laughs> κορμούς που φτάνουν σε ένα λιμάνι και στο λιμάνι της Αμβέρσας, εγώ είμαι Βελγίδα. Πού τα κρύβεις? Και επομένως... Όταν μπαίνουν αυτοί οι κορμοί με πλαστά πιστοποιητικά, ε, Αναρωτιέμαι κατά πόσον είναι αποτελεσματική η έλεγχη στα σύνορα. Μπορούν να ελέγξουν αυτά τα οποία εισάγονται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ελέγχουμε τους μετανάστες και δυσκολευόμαστε να ελέγξουμε την παράνομη ξυλία που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία να λειτουργούν λίγο καλύτερα όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Δεύτερον, δεν ε, συζητήσαμε πολύ ε, για τις έμεσες συνέπειες της αποψήλωσης, τις έμεσες μάλλον συνέπειες του εμπορίου για την αποψήλωση και στο θέμα της γεωργίας και μιλήσαμε για το φινικέ Δηλαδή θα μπορούσαμε ίσως να αναφερόμαστε και σε εντατική καλλιέργεια σόγιας ή ε, εντατική κτηνοτροφία. Και νομίζω ότι οι εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε και υπογράφουμε είναι ενδιαφέροντα εργαλεία για να μπορέσουμε να ε, δούμε πόσο επιταχύνεται αυτό το φαινόμενο της αποψήλωσης. Διότι αν έχουμε ενίσχυση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον πληθυσμό να διαχειρίζεται καλύτερα τα θέματα. Και από την άλλη, μέσω των εμπορικών συμφωνιών ε, δείχνουμε προτίμηση σε εντατικέ καλλιέργειε και εντατική κλινοκτροφία που καταστρέφουν τη γη και επομένω ο πληθυσμό δεν έχει ε, κανένα συμφέρον να κάνει μια βιώσιμη καλλιέργεια, αλλά προτιμάει να την πουλήσει. Διαπιστώνουμε ότι από τη μια έχουμε ε, μέτρα για να ενισχύσουμε το βιώσιμη ε, γεωργία και από την άλλη έχουμε μέτρα εμπορία που δεν ε, σέβονται καθόλου αυτή τη βιωσιμότητα. Επομένω, το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά σε αυτέ τι συμφωνίε. Και άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο θέμα αυτό, να υπενθυμίσω ότι είχε γνωμοδοτήσει για τη Σιγκαπούρη, και λέει σαφέστατα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνει το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης σε αυτές τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και έχει τη δυνατότητα να στείλει μια συμφωνία εάν δεν υπάρχει σεβασμός αυτών των υποχρεώσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Επομένως δεν είναι ε, βέβαιο ότι είναι πολιτικό το θέμα. Είναι ε, νομική η θέση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας το επιβάλλει. Και εγώ λοιπόν νομίζω ότι όταν μας επιβάλλει κάτι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καλό θα ήταν εμείς ως υπεύθυνοι πολιτικοί να σεβόμαστε την άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κάτι τελευταίο. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγαπά πολύ τις εθελοντικές συμφωνίες και ξέρω ότι δίνει μάχη για τις ε, υποχρεωτικές συμφωνίες. Αλλά όταν σε κάτι εθελοντικό ε, γνωρίζουμε ότι οι πολυεθνικές έχουν δεσμευτεί σε εθελοντικό επίπεδο να δημοσιεύουν την προέλευση του φινικέλου που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους. Και δεσμεύτηκαν ε, μέχρι το 2020 να δημοσιεύουν ε, όλη την προέλευση του φινικελαίου. Και τώρα ακούω από επιχειρήσεις όπως η Pepsi-Cola, η Kellogg's, η Johnson Johnson και θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλες, που είναι επιχειρήσεις που ε, έχουν μεγάλη δραστηριότητα στην Ευρώπη και λένε ότι δεν αναφέρουν την ε, χώρα προέλευσης του φινικελαίου. Ουσιαστικά λοιπόν επειδή είναι θελοντικά ε, θα πρέπει να τα περιορίσουμε και ότι όταν υπάρχουν πολυεθνικές που δεσμεύονται να κάνουν κάτι και τελικά δεν το κάνουν θα πρέπει να λάβουμε μέτρα πολύ πιο περιοριστικά, υποχρεωτικά για να μπορέσουμε να σεβαστούμε αφενός τους Ευρωπαίους καταναλωτές που θέλουν να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων και από την άλλη τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρόθεσμη για τροπολογίες είναι 23η Μαρτίου, μία η ώρα. Και θα εγκρίνουμε την γνωμοδότηση στην επόμενη συνεδρία μας τον Απρίλιο. Περνάμε λοιπόν τώρα σημείο 16 και πριν ψηφίσουμε να συγχαρώ την κυρία Ανίκα Γκρίνεμ που χτες το βράδυ βραβεύθηκε ε, χτες το βράδυ βραβεύτηκε ως βουλευτής της χρονιάς σε θέματα εμπορίου από το περιοδικό Κοινοβουλευτικός. Συγχαρητήρια. Οπότε πρώτη ψηφοφορία. Αφορά την συζήτηση που είχαμε την έκθεση της κυρίας Μπεγκίν. Λοιπόν, κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Πάρτε τις κάρτες σας λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας όλα μια χαρά ψηφίσουμε λοιπόν τώρα το σημείο 16 ε, επιστολές ε, προς την Νορβηγία κτλ έκθεση Μπεγκίν άρχιτε η ψηφοφορία Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Σημείο 17. Προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για περιοριστικά μέτρα για την Κρυμαία και τη Σεβαστούπολη. Άρχεται η ψηφοφορία. και πέρας. Εγκρίνεται. Σημείο 18. Πρώτη έκθεση του νέου συναδέλφου Έλση Κατάινεν για, της κυρίας Έλση Κατάινεν για την ε, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Ε, μόλις κατέφθασε για να ψηφίσει την έκθεσή της. Ωραία. Και πέρας ε, εγκρίνεται συγχαρητήρια λοιπόν για την έκθεσή σας. Αυτά με τις ψηφοφορίες τελειώσαμε. Ακολουθεί διάλειμμα λίγων λεπτών μέχρι να έρθει η Επίτροπος προσγειώθηκε στις ε, Βρυξέλλες ε, και κατευθύνεται τάχιστα προς το Κοινοβούλιο. 10-15 λεπτά, 20 διάλειμμα και κάνω μισά ώρα. Υπότιτλοι So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι. <laughs> and, uh, ε, τελείωσε το διάλειμμα. Wonderful looking. Έχω εδώ πέρα την ε, επειδή επίτροπο που ήρθε από την Ουάσιγκτον, ε, ε, ε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα αρχίσουμε τον ε, διαστομένο διάλογο με την ε, Επίτροπό μας, αρμόδια για τα εμπορικά θέματα. Ε, θα έχουμε εμεί κατά νου το πρόγραμμα εργασίας για το 2018, φυσικά και καυτά ζητήματα που συζητήσαμε και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Οι σχέσεις μας με Τσίπα και κάποια άλλα ζητήματα. 15-20 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητέ Μπέρντ, αξιότιμοι βουλευτέ. Ε, Κυρίε και κύριοι, καλημέρα. Ναι, είμαστε εδώ στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου. Ο στόχο είναι να συζητήσουμε τα πεπραγμένα Ε, στο τομέα του εμπορίου έγιναν πολλά ε, φέτος ε, διάφορες εμπορικές συμφωνίες και πολλές ενίκες κατά του προστατευτισμού αλλά και πολλές απώλειες, πολλές ήτες. Θα σας πούμε τι έχουμε κάνει, σε ποιο σημείο είμαστε και τι έπεται και φυσικά θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας συμφωνία με τον ε, Καναδά, η πλέον φιλόδοξη εμπορική συμφωνία με τον ε, Καναδά που έχει αρχίσει να ε, εφαρμόζεται, χαμηλέ τιμέ για του καταναλωτέ. μείωση δασμών, βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα και διατηρούμε παρόλα αυτά τα πρότυπα μα. Μετά από λίγες εβδομάδες οριστικοποιήθηκαν οι διαπραγματευτικέ μα συνομιλίε με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι ο έκτος μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο τη Ευρωπαϊκής και μία από τι μεγαλύτερε οικονομίε του κόσμου. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ωφέλη. Συμφωνία με το Βιετνάμ προστίθεται στον κατάλογο να θυμόμαστε, είναι σημαντικό, πως δεν είναι μόνο οικονομικές αυτές ε, όλες οι συμφωνίες. Είναι συμμαχίες στρατηγικού χαρακτήρα που οικοδομούμε με τους για να καθοδηγήσουμε την παγκοσμιοποίηση, να υπερασπιστούμε το ε, ανοιχτό εμπόριο και να συμφωνήσουμε για κανόνες που είναι δίκαιοι και μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από όλους. Ε, πρόκειται για διαφορετικές συμφωνίες που ανταποκρίνονται στις αξίες μας, στον ΟΣΑ, στη διευπουργική Αμερική, στο βλέπουμε ε, ότι οι εταίροι, κάποιοι αποχωρούν, κάποιοι νέοι έρχονται, αλλά πάντως ε, η γενικότερη τάση είναι ότι υπερασπίζονται το δίκαιο και ελεύθερο εμπόριο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά την ε, ήττα στο Μπένο Άρε με τον τελευταίο κύριο των διαπραγματεύσεων. Το πολυμερές σύστημα έχει αποτελματωθεί και εργαζόμαστε σκληρά για, να το, για την απεμπλοκή του και έχουμε ένα ηγετικό ρόλο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ εξελίξεις. Ε, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνησε ε, στην ε, απόφασή της τα θέμα περιμικτού καθεστώτος. Έχουμε πολύ σημαντική ανάλυση για το GSP, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Έχουμε κάνει άλματα υπέρ της διαφάνειας από το Σεπτέμβρη και μετά. Ε, δημοσιεύουμε όλα τα σχέδια οδηγία εμπορικού χαρακτήρα και τα στέλνουμε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αρχίσει νωρίτερα η συμφωνία και εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς ε, στη, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων προτού εγκριθούν οι οδηγίες ενημερώνουμε το κοινό για την ε, πορεία των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια του γύρω του διαπραγματευτικού και σχετικό υλικό, κοινωνία των πολιτών, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορές όπως κάναμε και για τη Σέτα. Ε, τώρα έχουμε και μια συμβουλευτική ομάδα για την κοινωνία των πολιτών. Ε, βλέπετε ε, συγκεκριμένα αυτά παραδείγματα πώς μεταφράζεται η πρόθεσή μας σε δράση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τη συμφωνία με τον Καναδά. Έχουμε χαρτογραφήσει τα επόμενα βήματα, τρεις τομείς για την εφαρμογή, θεσμικό πλαίσιο, αεραβάθμιση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων για την βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες προκατακτικές συνεδριάσεις και ε, προώθηση ε, του Δικαστηρίου Διευθέτησης Διαφορών. Ε, θα είναι χρονοβόρια η διαδικασία της επικύρωσης, αλλά Αν δούνε αυτά αποτελέσματα κράτη-μέλη θα επιταχυνθεί η διαδικασία. Για την συμφωνία τη Ιαπωνία από νομική πλευρά θα έχουμε χτενίσει το κείμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το εγκρίνει το κείμενο και θα σα το στείλει στι 17 Απριλίου. Θα σα το στείλουμε και θα το στείλουμε και στο Συμβούλιο. Το μπαλάκι θα είναι στο δικό σα γήπεδο και ελπίζουμε ε, να ε, δουλέψετε ταχύτατα όπω και εμεί. Ε, πλησιάζουμε το κλείσμα τη συμφωνία με το Μερκοσούρ και το Μεξικό. Είναι εντατικέ οι διαπραγματεύσει. είναι ιδιαίτερα σημαντικέ συμφωνίε για μας. Φυσικά όμως ε, ε, δεν ε, θυσιάζουμε τα πρότυπα μα για να επιταχύνουμε την επίτευξη τη συμφωνία, αλλά κάνουμε πάρα πολύ σημαντικέ προσπάθειε και πολύ σύντομα, σε επόμενε εβδομάδε στον επόμενο μήνα, ελπίζουμε να καταλήξουμε. Ε, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ε, συζητούμε Διαπραγματευόμαστε για τις εντολές ε, και ελπίζουμε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πριν το καλοκαίρι αν εγκρίνουν και εκείνες οι διαπραγματευτικές εντολές. Ε, η σχέση μας με την Κίνα είναι περίπλοκη αυτή η σχέση. Ε, πολύ βασικό εμπορικό εταιρό, αλλά για το εμπόριο και για την οικονομία έχουμε πολύ διαφορετικές ε, ε, απόψει και δεν βλέπουμε πάντοτε ή όρου ανταγωνισμού για τι εξαγωγικέ αγορέ μα ή για τι συνθήκε που ισχύουν για τι επιχειρήσει μα πάντα. Οπότε θα συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει για την αμοιβαιότητα, για την ισότητα των όρων ανταγωνισμού, για την υπερδυναμικότητα, για την πρόσβαση στην αγορά. Όλα αυτά θα είναι θέματα εστίαση ε, στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα σε τριμερή συνεργασία που αρχίσαμε επίσης ε, με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Τα ίδια θέματα μας αποσχολήσουν όπως είπε και ο Πρόεδρος. Ε, μόλις έφτασα πριν από δύο ώρες από την Ουάσιγκτον ε, ε, φέτος ε, άλλαξαν πορεία προς την εμπορική πολιτική. Δυστυχώς ε, απομακρύνονται από τον ΠΟΕ, δεν διορίζουν νέους δικαστές. Αυτό απειλεί ολόκληρο το πολυμερές σύστημα και δεν επικεντρώνονται στις διατλαντικές σχέσεις τόσο πολύ όσο στις σχέσεις με την Κίνα. Επιθετική, επιθετικότερη χρήση των οργάνων υπεράσπισης του εμπορίου και παρά το αρνητικό πλαίσιο μπορέσαμε με οικοδομητικό τρόπο να να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Ε, Παραδείγματο χάρη στι τριμερεί ε, συνεδριάσει για την ε, υπερδυναμικότητα, συνεχίζουμε τι συζητήσει. Όπω ξέρετε, για το αλουμίνιο και για το χάλιβα, στι 8 Μαρτίου εξήγηλε η κυβέρνηση Τραμπ τι κυρώσει βάσει τη νομοθεσία 232 για θέματα εθνική ασφάλεια. Όπω γνωρίζουμε όλοι, αυτό είναι ασύμβατο με την απόφαση του ΠΟΕ για τα συγκεκριμένα προϊόντα και Σίγουρα εμείς δεν πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτό, είμαστε φίλοι και εταιροί και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούμε απειλή ε, κατά της ε, ε, εθνικής ασφάλειας. εντατικά συνεργαζόμαστε με τον πρέσβη Αιτάιζερ και με τον Υπουργό Εξωτερικών Ρώσο και ε, πριν από λίγες εβδομάδες ε, στην κοινή συνεδρία και με την Ιαπωνία ε, αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα της υπερδυναμικότητας κυρίως στην παραγωγή στην Κίνα και αυτό το πρόβλημα ε, προέρχεται από την Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει, η βιομηχανία μας ε, υποφέρουν, ε, έχουν πληγεί από αυτό το φαινόμενο στον τομέα του Χάλιβα. Έχουμε τροποποιήσει τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για την υπεράσπιση του εμπορίου με τη δική σας βοήθεια στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το εμπόριο στα προϊόντα χαλιβουργίας. Έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα συνεχίζουμε τον αγώνα. Έχουμε ε, κάποια συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, δηλαδή έχουν χρησιμοποιήσει κριτήρια γιατί ε, θα έπρεπε να μας αποκλείσουν από αυτή την διαδικασία και το βασικό καταλητικότερο επιχείρημά μας ε, ήταν ότι θα μιλάμε με μία φωνή. θα παραμείνουμε ενωμένοι με το, συζητήσαμε το θέμα με τον κύριο Ρώσο και είπε ότι ε, θα ε, προτείνει στον πρόεδρο Τραμπ να ε, μας αποκλείσει από τις κυρώσεις. Σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνει τις εξαγγελίες του. Ελπίζουμε να συμπεριληφθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, εν πάση θα κάνει τη σύστασή του ο κύριος αλλά αποφασίζει ο κύριος Τραμπ. Ε, σήμερα το απόγευμα θα το εξαγγείλει ο πρόεδρος Θεόμ και ελπίζουμε να εξαιρεθεί η ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε θα συσταθεί η ομάδα εργασίας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ε, γενικότερα για εμπορικά ζητήματα ότι έχει σχέση με την ε, προστασία των επενδύσεων και θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Είπαμε υπερδυναμικότητα παραγωγής, ε, θέματα χαλιβουργίας και ούτω καθεξής. Παραλλήλου και δηλώνουμε ξεκάθαρα, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι αν ε, μας επιβάλλουν αυτούς τους ε, δασμούς θα αναλάβουμε δράση και θα ε, κινηθούμε αντίον τους στα πλαίσια του ΠΟΕ, όπως και άλλες χώρες. Συνεχίζουμε τη δουλειά για τις ειδικλείδες ασφαλείας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι πλήγει η βιομηχανία, η χαλιβουργία για λόγω της ψυχολογίας της αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν να επανισορροπήσουμε τα μέτρα. Είδα τον τελευταίο κατάλογο που δημοσιεύσαμε το... την Παρασκευή και συνεχίσουμε τώρα την... το διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς ε, στα κράτη-μέλη. Δεν είναι σαφής η διαδικασία. Υπάρχουν ερωτηματικά, πρέπει να διαλευκάνουμε κάποια ζητήματα και είπαμε ότι το απόγευμα ή το βράδυ, ευρωπαϊκή ώρα, Έχουμε την εξαγγελία από πλευράς του Πρόεδρου Τραμπ και ε, θα σύντομα θα έρθουμε σε επαφή με του ομοτήμου μα για τη σύσταση αυτή τη ομάδα εργασία, να δούμε πώ θα διαμορφωθεί. Ξέρω, θα έχετε πολλές ε, ερωτήσει γι' αυτό, αλλά θέλω να ολοκληρώσω τώρα την εικόνα για όλα τα εμπορικά ζητήματα και μετά θα τα δούμε. Ε, ε, με τη χιλή, διμερεί διαπραγματεύσει και εκεί έχουμε σημειώσει πρόοδο. σε κάποιου τομεί ακόμη δεν έχουμε λήξει συμφωνία. το δουλεύουμε όμω, όπω παραδείγματο χάρη, με τα ρυθμισμένο σύστημα ISDS για διαφορών Λοιπόν, ε, ε, έγιναν εκλογές όπως ξέρετε και καθυστερήσαμε, αλλά νομίζω το Μάιο θα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι για το εμπόριο και την ισότητα των δύο φίλων μπορούμε να κάνουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα μέσα στα πλαίσια της Θελοντικής Συμφωνίας Ελευθέρου μπορούμε την Χιλή. γενικότερα με τους εταίρους μας νομίζω ότι υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη συμφωνία ότι το εμπόριο συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουν, είναι προοδευτικοί, θέλουν να συνδέσουν το εμπόριο με τη βιωσιμότητα και με τις αρχές ε, των οποίων περαμεινόμαστε ή να συνδέσουν το εμπόριο με συνθήκε συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι αυτές ακριβώς είναι και οι αξίες που θέλουμε εμείς να μεταδίδουμε μέσα από τις συμφωνίες, ε, ε, συνθήκες εργασίας, δικαιώματα εργασίας ε, ε, βιωσιμότητα περιβάλλον. Ε, τώρα έχουμε κάνει προτάσεις για αναβίωση ε, της ε, μας σύνδεση του εμπορίου με τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από 15 πολύ συγκεκριμένες ε, δράσεις ενίσχυση της συνεργασίας, δυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα, δημοσίευση, διαφάνεια. Ε, αυτές είναι οι απαντήσεις που δίνουμε στις ε, ελλείψεις που εντοπίζουμε σε σχέση με την κατάσταση όπως έχει τώρα και προωθούμε αυτές τις δράσεις. Ξέρετε ότι αλλάζει ο κόσμος και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διεξάγουμε τις εμπορικές μας συναλλαγές και γι' αυτό για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και όταν δεν ακολουθούνται οι κανόνες από τους εταίρους μας έχουμε τροποποιήσει τα μέσα προστασίας μας για να έχουμε ταχύτερη αντίδραση για να καταπολεμήσουμε τη στρέβλωση υπέρ των επιχειρήσεών μας. Έτσι έχουμε ένα δικαιότερο εμπορικό σύστημα και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί εργαστήκατε σκληρά μαζί μας το Δεκέμβρη καταλήξαμε σε μια ιδιαίτερα ισορροπημένη συμφωνία. Επικείμενες ε, προκλήσεις, ε, ε, στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία ποιοι ενωσιακούς επενδυτές που καλωσορίζουμε τις επενδύσεις αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε ότι πρόκειται για επιδοτούμενες επιχειρήσεις που στηρίζονται άμεσα από κυβερνήσεις κάποιων κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για μεταβίβαση τεχνογνωσίας, ε, θέματα ιδιοκτησίας. Ε, θα πρέπει λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλάβουμε τι ακριβώς ε, συμβαίνει, να έχουμε τη σφαιρικότερη εικόνα και χαίρομαι που θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Προύστης. Η εμπορική πολιτική της Ένωσης πρέπει να συνεισφέρει στην ασφάλεια της υπηρού μα αλλά και στην ανθρώπινη ασφαλεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Χαίρομαστε λοιπόν για το ότι θέλετε να παρακολουθούμε την χρήση και κατάχρηση των προϊόντων διπλής χρήσης, ειδικά όταν μιλάμε για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν θα συνεισφέρουμε σε έναν ασφαλέστερο κόσμο, όπως άλλωστε και η Παγκόσμια Συμμαχία κατά των βασανιστήριων και της θανατικής ποινή, που έχει αυτή τη στιγμή 58 χώρες ε, συμβαλόμενες. Και βεβαίως ε, συνεργαζόμαστε και σε διμερές επίπεδο, αλλά ε, είμαστε πάρα πολύ ε, δεσμευμένοι στο πολυμερές σύστημα. Είδαμε τις συζητήσεις των Buenos Aires, ε, τις διαπραγματεύσεις και τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Για να απαντήσουμε σε αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα και να συνεργαστούμε με άλλους. Θέλουμε να διατηρήσουμε τον μηχανισμό αυτό επίλυσης διαφορών και το μηχανισμό εφέσεων. Θέλουμε επίσης να αναζητήσουμε εναλλακτικέ προσεγγίσεις για να ξεμπλοκάρει ο ΠΟΕ με διμερείς επαφές και θα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ζητήματα όπου υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον, Παραδείγματος χάρη στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα προωθήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά γεγονό είναι ότι ο ΠΟΕ χρειάζεται κάποια ηγεσία, κάποια μεταρρύθμιση και σκοπεύουμε να ε, καταφέρουμε να λειτουργήσει. Είναι σημαντικός για το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Για αυτό τον λόγο αποδίδουμε μεγάλη σημασία στο πολυμερές ε, δικαστήριο επενδύσεων. Ε, προχωράμε σε αυτό το μέτωπο. Το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει διαπραγματευτικές οδηγίες, κάτι το θετικό γιατί το παλιό σύστημα ε, είναι πλέον ξεπερασμένο. Υπήρχε μια πρώτη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, η επόμενη θα λάβει χώρα τον Απρίλιο. Σχηματίζουμε λοιπόν συμμαχίες ε, και αναμένουμε θετικές εξελίξεις. Ξέρω πως αυτό είναι σημαντικό για πολλούς από εσάς. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα ζητήματα που μας απασχολούν. Ε, το Brexit επίσης ε, προχωράει. Ε, για, θα μας επηρεάσει. Πρέπει να σκεφτούμε το εμπόριο και στην δική μας την ε, περιοχή. Και βεβαίω αυτό θα επηρεάσει το πώς ε, λειτουργούμε, το πώς εμπορευόμαστε, αλλά νομίζουμε ότι έχουμε τα εργαλεία και τις πολιτικές να το δούμε αυτό φτιάχνουμε μια μεγάλη ομάδα φίλων και συμμάχων, η εμπορική πολιτική μας νομίζω μπορεί να ανταποκριθεί. Ο κόσμος ε, στρέφεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεργασία και τώρα μπαίνουμε αυτό και βεβαίως ε, συνεργαζόμαστε μαζί με την ΙΝΤΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και με αυτά τα ολίγα σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ε, και αναμένω να ακούσω τι έχετε να πείτε. Ωραιότατα, σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Θα δώσω τον λόγο πρώτα απ' όλα στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων για τρία λεπτά ο καθένας. Η Χοντελίβε από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ε, σας καλωσορίζω και βεβαίως φαντάζομαι θα είστε πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένοι βλέπετε κάποια ε, δυνατότητα, ε, ίσως είμαι πολύ αισιόδοξη, η κρίση αυτή που ζούμε τώρα με την κυβέρνηση Τραμπ και την κατάσταση που γνωρίζουμε να αποτελεί και μια ευκαιρία να έχουμε κάποια συμφωνία, όχι την TTIP, με κάποιο άλλο όνομα, να ξαναξεκινήσει λοιπόν μια διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς. Έχω διαβάσει διάφορα σχετικά. Το ένα είναι αυτό. αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η άλλη αφορά τη μεταρρυθμίση του ΠΟΕ. Θέλουμε να σκεφτόμαστε πολυμερός, όχι μόνο να σκεφτόμαστε, αλλά και να δρούμε έτσι. Έχετε μια πιο συγκεκριμένη άποψη για το τι μορφή θα μπορούσε να έχει μια τέτοια μεταρρύθμιση. Το τρίτο θέμα. Βεβαίω και εσείς και το ΕΛΚ ε, είμαστε υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης ε, κτλ. και είμαι σίγουρος, αλλά μήπως ε, ακριβώ ε, παραφορτώνουμε πολλά πράγματα στους εμπορικούς μας εταίρους και ζητάμε τα πάντα. Μήπως υπάρχει κάπως η δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια ισορροπία Επόμενη ερώτηση και τελειώνω επιτέλους. Προστασία των επενδύσεων, πάντα το ίδιο θέμα. Θέλουμε ένα πολυμερές ε, δικαστήριο, αλλά κράτη δεν το θέλουν. Υπάρχει κάποιο σχέδιο Β που έχετε προετοιμάσει ή κάποια ενδιάμεση λύση. Και η τελευταία τελευταία ερώτηση κάτι το οποίο με αφορά προσωπικά. Υπάρχει κάποιο όριο στις δυνατότητες εμπορίου. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε μια διαφορετική ανάπτυξη. Είναι τελείως προσωπική ε, η ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω, ίσως έχετε σκεφτεί κάτι, ίσως όχι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Αρένα λοιπόν για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς η πρώτη ερώτηση βάσει και των συζητήσεων που είχατε στη Washington ε, είμαστε πριν από την εφαρμογή των δασμών ε, για το χάλιβα και το αλουμίνιο από πλευρά των ΗΠΑ και τι αίσθηση έχετε μετά τη συζήτηση εχθέ. Ε, εχθέ ο κ. Δεμαρτή έλεγε ότι δεν συζητάμε υποπίεση, αλλά το θέμα είναι τι νεότερα έχουμε από τι ΗΠΑ για αυτά τα προστατευτικά μέτρα για το χάλιβα και το αλουμίνιο. Επίση, για τον Καναδά. Μα είπατε ότι ε, φτάνετε στη ρήτρα αναθεώρηση και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα του κεφαλαίου της βιώσιμης ανάπτυξης. Ποιες είναι οι βελτιώσεις που ε, είστε διατεθειμένοι και εσείς και οι εταίροι να κάνετε. Ξέρετε ότι ο Καναδάς ε, είχε μια οπτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη με κυρώσεις. Πού βρισκόμαστε σε αυτή τη συζήτηση με τον Καναδά. Ε, επόμενη ερώτηση. Η άποψη της Σιγκαπούρης. Γιατί η Σιγκαπούρη... Ε, βάσει τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να συμπεριλάβει και στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στην ε, εμπορική πολιτική και μια πολιτική ελευθέρων συναλλαγών μπορεί να ανασταλεί στην περίπτωση που η βιώσιμη ανάπτυξη δεν γίνεται σεβαστή και οι διατάξεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν γίνονται σεβαστές. Πώς ε, θα ερμηνεύσετε αυτή την ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην περίπτωση της Σιγκαπούρη για όλες τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Τέταρτον, και πάλι για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπήρξε μια γνωμοδότηση ή μάλλον απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ε, Γεωργική και Αλληλευτική Συμφωνία με το Μαρόκο. Ε, πού βρίσκεστε, ξέρω ότι υπάρχουν ε, διαπραγματεύσεις, εκπνέει η Συμφωνία τον Ιούλιο και επομένω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. 5. Συμφωνία Μερκοσούρ. Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας ε, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Εσείς ε, πώς ανταποκρίνεστε σε αυτές τις ευαισθησίες του γεωργικού τομέα στα πλαίσια της συμφωνίας Μερκοσούρ. Για τη συμφωνία για την Ιαπωνία ε, είπατε ένα-δυο πράγματα και κάναμε μια συζήτηση πριν σας ακούσουμε για το θέμα της αποψήλωσης των δασών. Γνωρίζουμε ότι η Ιαπωνία είναι ο τέταρτος παγκόσμιος εισαγωγέας ξυλίας ε, και μεταποιημένης ξυλίας και γνωρίζουμε επίσης <laughs> ότι οι συμφωνίες είναι εθελοντικές με την Ιαπωνία όσον αφορά τα πιστοποιητικά ξυλίας. Πώς ε, θα προχωρήσετε για μια πιο ε, υποχρεωτική ρύθμιση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τι εθελοντικέ συμφωνίε που έχουμε με την Ιαπωνία και πώ θα τα συμφιλιώσετε αυτά τα δύο. Επίση, είχαμε την ε, πολυμερή συμφωνία επενδύσεων από πλευρά Συμβουλίου. Εσεί ε, πώ θα υλοποιήσετε την εντολή που σα δόθηκε από το Συμβούλιο για το θέμα τη ε, σύσταση του ε, πολυμερούς δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ από πλευρά ECR η Emma clarking. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις προσπάθειες που κάνατε για να ε, δώσετε αποτελέσματα στα θέματα εμπορίου και κυρίως τη γρήγορη αντίδρασή σας ε, για την ε, στάση των ΗΠΑ. Ήταν εντυπωσιακά αυτά που κάνατε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ανεπίσημο έγγραφο στο non-paper για την εφαρμογή των κεφαλαίων TST. Ευπρόσδεκτη πρόταση από πλευρά ECR και χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προκύπτει σε πιέσει για μια προσέγγιση βάση κυρώσεων για το θέμα αυτό. Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσει θα βοηθήσει τη βιωσιμότητα, ενώ το αν το επεξεργαστούμε ε, θα έχουμε αποτελέσματα. Το έγγραφο αναφέρεται σε μια προσέγγιση αναχώρα. Είναι η καλύτερη προσέγγιση αυτή, το να έχουμε διαφορετικά κεφάλαια σε κάθε χώρα ή θα έπρεπε να έχουμε μια πολυμερή συμφωνία για τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω, όπω για παράδειγμα συμφωνίες των Παρισίων, αντίστοιχο του Διεθνου Γραφείου Εργασία κλπ. Ε, και επίση, για τη στρατηγική για το εμπόριο είπαμε ότι θα εξετάσουμε και ε, διαπραγματεύσει για επενδύσεων με την Ταϊβάν και την Νότια Κορέα. Έχετε ακόμα αυτή την φιλοδοξία και υπάρχουν κάποια σχέδια για αξιολόγηση επιπτώσεων για μελλοντικέ τέτοιε συμφωνίε επενδύσεων. Αναφερόμαστε πολύ για το χρονοδιάγραμμα για την Ιαπωνία και το Σιγκαπούρη. Ε, θα γίνουν αυτά στη διάρκεια αυτή τη εντολή ή θα καθυστερήσουν. Και τέλο. Υπάρχουν και οδηγίες διαπραγμάτευσης οι οποίες ε, δημοσιεύτηκαν για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Πότε θα δούμε συμφωνία στο Συμβούλιο για την εντολή. Θα ήθελα να γνωρίζω, νομίζω και οι υπόλοιποι. Με χαρά ακούω ότι προετοιμάζεστε για το Brexit. και ξεκινάτε τι διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσει συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε εγώ είτε η ομάδα μου, είμαστε στη διάθεσή σας και είμαστε και έτοιμοι. Ευχαριστώ πολύ. Η Χάιντι Χάουταλα αντικαθιστά το Γιάννη Ζαντό από τους Πρασίδνους. Η φιλελεύθερη μετά. Ναι, εντάξει, να υποκύψω στους πρασίνους, ε, πρόεδρος. Ναι, η Μαρία Τεσχάκε ε, για τους, πρασί... για τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πολύ. Είναι νωρίς για όλους. Καλημέρα κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε να μας ενημερώσετε ε, άρτια φιχθήσα μόλις βγήκατε από το και μάλιστα μετά από τόσες δύσκολες διαπραγματεύσεις έχετε όλοι μας την υποστήριξη και ελπίζω να μπορέσουμε να είμαστε ενωμένοι και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Εξετάζοντα την προηγούμενη χρονιά, έχουμε πολύ σημαντικά διδάγματα. Τα θίξατε τα περισσότερα από αυτά και ελπίζω να μα βοηθήσουν και στη συνέχεια. Νομίζω ότι έχει γίνει μια δραματική αλλαγή στον τόνο τη συζήτηση. Οι εξελίξει ε, με τον Τραμπ και τον Brexit ήταν αφύπνιση για όσοι το χρειαζόντουσαν και νομίζω ότι φαίνεται ότι στην Ευρώπη έχουν όλοι αντιληφθεί ότι χρειαζόμαστε να αναλάβουμε τα ενία και να αναπτύξουμε εταιρικέ σχέσεις και χαίρομαι που βλέπω ότι εσεί αναλαμβάνετε αυτό το ρόλο και βρίσκεστε στο πιδάλιο. Ίσως θα προσέξετε επίση ότι την προηγούμενη εβδομάδα στη συζήτηση στο Στρασβούργο υπήρχε ανανεωμένη εκτίμηση από κάποιους συναδέλφους οι οποίοι ε, αμφισβητούσαν το σύστημα εμπορίου βάση κανόνων με κάθε ευκαιρία και τώρα φαίνεται να το εκτιμούν γιατί δεν θέλουν να βρεθούν ε, στο πεδίο του Τραμπ ε, όσον αφορά το εμπόριο και σίγουρα εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να βρεθούμε εκεί. Σίγουρα διακυβεύονται πολλά και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία πάρα πολύ προσεκτικά. Και βεβαίω ε, το να έχουμε στενότερη συνεργασία με βασικού εταίρου που μοιράζονται τι αξίε μα όπω ο Καναδά, το Μεξικό, η Ιαπωνία είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε νέε συμμαχίε όπω αναφέρεται το Μερκοσούρ είναι πολύ σημαντικό αλλά και νέους τομείς εμπορίου, ψηφιακού εμπορίου ε, έλεγχος των επενδύσεων ε, σε δυνητικά κρίσιμους ε, τομείς και ο κανονισμός για τα προϊόντα της χρήσης. Μία ερώτηση γιατί μόλις ήρθατε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μας αποσχολούν πολλά. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαίρεση, θα αμφισβητήσετε για λόγους αρχής την επίκληση ε, λόγων ε, εθνικής ασφάλειας. Ε, φυσικά όλοι θα ήταν ιδιαίτερως ικανοποιημένοι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση λάβει την εξαίρεση που της αξίζει, αλλά το επιχείρημα της εθνικής ασφάλειας είναι προβληματικό. Και φαίνεται ότι υπάρχει σύγχυση και σε υψηλό πολιτικό επίπεδο για την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί να δραστηριοποιείται συνολικά. Άκουσα από κάποιους, δεν θα πω ποιους, χθες, ότι αν μια τρίτη χώρα προσφέρει ειδική μεταχείριση σε ένα κράτος μέλος, το κράτος μέλος μπορεί να τη δεχτεί, ενώ δεν μπορεί να δεσμευτεί σε εξαιρετικά μέτρα εμπορίου ε, με τρίτες χώρες. Ίσως θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, κυρίως με τις χώρες μέλη, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που θεωρούν ότι μπορεί να λάβουν εξαίρεση ή ειδική μεταχείριση, όπως ε, ε, ανέφερε ο κύριος Κραμπ και, ε, Τραμπ και νομίζω ότι το να υπονομεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή θα είναι εις βάρος μας και για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο είναι ακόμα μέλος. Και κάποιοι αναφέρουν ότι αυτό το δραματικό ε, ναβύρ στι εμπορικέ σχέσει με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού μπορεί να οδηγήσει σε ανανεωμένε διαπραγματεύσει. Για μένα αυτά είναι φρούδε ελπίδε. Ε, σω θα μπορούσατε να μα πείτε εσεί αν υπάρχει περιθώριο και αν υπάρχει οτιδήποτε επικοδομητικό, διότι μόλι επιστρέψατε από εκεί. Ευχαριστώ και τώρα για του πρασίνου. Η κυρία Χάουταλα, ευχαριστώ. Τώρα πρόσεξα ότι η ομάδα μου είναι κάπω μεγαλύτερη από την ΚΟΕ. Με πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, ευχαριστώ που ήρθατε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για το ότι δημοσίευσατε την διαπραγματευτική σας εντολή για το πολυμερές ε, επενδυτικό δικαστήριο και νομίζω ότι μπορείτε τώρα να πείστε και το Συμβούλιο να κάνει το ίδιο. Αλλά η ομάδα μου απογοητεύτηκε με το περιεχόμενο της εντολής γιατί περιμέναμε τουλάχιστον κάποια διαδικαστικά δικαιώματα να έχουν πρόσθεθει για να ενισχυθούν τα δικαιώματα των κρατών ή άλλων μερών. Γιατί λοιπόν δεν προτείνατε παραδείγματο χάρη το δικαίωμα αντιπροσφυγών ως ε, ε, ένα ελάχιστο βήμα αντιστάθμισης των δικαιωμάτων των επενδυτών. Σε σχέση με αυτό, προσφάτως, υπήρχε μια απόφαση του ΔΕΚ για μια συμφωνία μεταξύ Ολλανδίας και Σλοβακίας, βεβαίως δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα σε σχέση με το σύστημα του επενδυτικού δικαστηρίου στην ΣΥΤΑ, αλλά η υπηρεσία σας πώς αναλύουν την απόφαση του δικαστηρίου ε, όσον αφορά την ε, Ολλανδία, καθώς ε, η απόφαση ήταν ότι δεν συμφωνεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με την απόφαση που αναμένουμε για το μηχανισμό της ΣΥΤΑ. Η άλλη μου ερώτηση βεβαίω αφορά το εμπόριο και τις βιώσιμες σχέσεις. Συγκεκριμένα, όπως ξέρετε, οι χώρες που καλλιεργούν φινικέλιο ανησυχούν ιδιαίτερα στο κοινοβούλιο, γιατί στη σχετική οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουμε πει ότι το φινικέλιο πλέον δεν ε, πρέπει να περιλαμβάνεται στους μηχανισμούς διπλής μέτρησης ε, ε, για την κλιματική αλλαγή. Και προφανώς ε, μπορεί να υπάρχουν κάποια ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο. Αλλά η θέση αυτή του Κοινοβουλίου να μην ευνοείται πλέον το φινικέλαιο μετά το 2021 είναι ένα σαφές μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο θέλει να πάρει στα σοβαρά τα... τις αρνητικές επιπτώσεις ε, του φινικελαίου και την αυξανόμενη ζήτηση για βιοκαύσιμα στην Ευρώπη. Πρέπει να βρεθεί κάποιο τρόπο για να καλέσουμε την Ινδονησία και άλλε χώρε να λάβουν κάποια μέτρα για να κάνουν κάτι για τις ανησυχίε μα, την αποδάσωση, αλλαγή χρήση γης, δικαιώματα αυτοχθόνων πληθυσμών. Μήπως έτσι μπορούμε να δούμε το ποια θα μπορούσε να είναι μια συνολική απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες για να συνεχιστεί το εμπόριο. Χέλμουτ Σόλτ για την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε που αμέσως μετά την προσγειώσή σας ήρθατε εδώ να μας ενημερώσετε για κάποια αποτελέσματα, αλλά βεβαίως και για να διατηρηθεί ο δομημένος διάλογος και βεβαίως ε, εντάξει ε, λυπούμε τώρα που είμαστε λιγότεροι από τους πράσινες αλλά οι συμφωνίες εξακολουθούν να ισχύουν ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία τα αποτελέσματα των συνομιλιών που είχατε στην Ουάσιγκτον στην ε, Επιτροπή Δημοσίων Οικονομικών. Ε, από ό,τι πληροφορήθηκα, σας είπαν εκεί ότι θέλουμε να αποφύγουμε έναν διατλαντικό εμπορικό πόλεμο. Ε, πρέπει να το βάλουμε σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Πρέπει να αποφύγουμε έναν εμπορικό πόλεμο γενικώ. Διότι οποιοδήποτε αποκλεισμό θα μπορούσε για κάποιες βιομηχανίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ε, ένα θετικό βήμα, αλλά εάν ε, έχουμε δασμούς στο χάλιβα από την Τουρκία, τη Λευκορωσία ή κάπου αλλού, θα κατευθυνθεί αυτός ο χάλιβας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να οργανωθεί μια γενική συζήτηση για την παραγωγή, για τις ποσοστώσεις και πρέπει να βρεθεί μια γενική λύση για να μειωθεί η υπερβολική παραγωγή, αλλά βεβαίως υπάρχουν και οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με αυτήν. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα δηλαδή, πώς θα πάμε στις πολυμερείς αυτές συζητήσεις για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Δεύτερη ερώτηση, αναφέρατε ότι θέλετε να δείτε τι θα γίνει Μερκοσούρ και του Μεξικού, το ανέφεραν και πολλοί συνάδελφοι, ότι οι προκλήσεις για τα γεωργικά είναι από τη δική μας ε, τη σκοπιά πολύ μακριά από εκεί που θα θέλαμε. Δεν βλέπουμε κάποιο όφελος για τους πολίτες της ε, χώρες που επηρεάζονται. Αλλά παίρνοντας σαν παράδειγμα το κεφάλαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας ε, για τις φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχουν παράγματι πολλές βιομηχανίες που παράγουν γενώσιμα, αλλά <coughs> και μήκυο ε, που λένε ότι η πρόσβαση των πολιτών στα φινά φάρμακα θα κινδυνεύσει με τις συμφωνίες αυτές. Και το ίδιο πρόβλημα τώρα θα προκύψει στο Μεξικό. Σκοπεύετε να προσαρμόσετε κάτι πώς σκοπεύετε να ξεπεράσετε τους φόβους των πολιτών. Τέλος, για την Κίνα. Είπατε, ναι, ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εμπορική συμφωνία. Πώς σκοπεύετε ακριβώ να βελτιώσετε την ικανότητά μας να καταλήξουμε σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα με τους ε, Κινέζους, λάμβανοντας υπόψη ακριβώς όπως είπατε, τις διαφορές ε, των οικονομιών. Ε, κύριος Ντάρτμοθ για το EFTD, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες της ομάδας μου που ήρθατε τόσο γρήγορα μετά από μια τόσο μεγάλη πτήση. Τα έκανα αυτά και εγώ όταν ήμουν 20 χρόνων. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να κάνω μια ερώτηση με στόχο να αποσπάσω πληροφορίες. Υπάρχει ένας τίτλος του Reuters που λέει «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει διαδικασία αντιπίνων κατά των δασμών των ΙΠΑ». Μετά από λίγες μέρες ε, η Washington Post λέει αντιπαράθεση για τον Χάλιβα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία πιέζουν ε, τις ε, σύμμαχες είπα για εξαίρεση. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικό σας, ε, η δική σας Γενική Διεύθυνση έχει ζητήσει εξαίρεση αντί για αντίπεινα και εάν έχετε αποφασίσει κάτι τέτοιο και δεν υπάρξει τελικά εξαίρεση σκοπεύετε να προβείτε σε αντίπεινα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές ήταν οι ερωτήσει μου. Μπορεί κάποιο άλλος να χρειαστεί τον χρόνο. Ωραιότατα. Τον λόγο έχει λοιπόν η κυρία Επίτροπος να απαντήσει στους συντονιστέ και μετά τελειώνει ο κατάλογος των ομιλητών. Έχουμε 10 βουλευτέ. Αν υπάρχει κάποιο άλλο. Όχι, ωραία κλείνει εδώ ο κατάλογος. Οι συνάδελφοι έχουν δύο λεπτά αφού τελειώσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες από τις ερωτήσεις ε, επαναλήφθηκαν, οπότε θα τις απαντήσω ε, μαζί. Για την ερώτησή σας, ε, κυρία, όχι, δεν βγάζουμε την δίτυπα από την κατάψυξη. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν την επόμενη εβδομάδα αλλά ο στόχος είναι να γίνει μια πολύ ευρύτερη συζήτηση για γενικά θέματα ενδιαφέροντας, ε, κάποια ε, στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αλλά και μια ευρύτερη συζήτηση εν γέννη. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε θα έρθουμε σε επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξαιρεθούμε βεβαίως, και ε, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό. Πάντα είμαστε διατεθειμένοι βεβαίως να συζητήσουμε. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο σημείων που μας ενοχλούν, ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας, όπου και για πάρα πολλά χρόνια ε, περιμένουμε πρόσβαση στις αμερικανικές αγορές για όλες τις χώρες μας, αλλά είναι πάρα πολύ περιορισμένοι και ε, αν είναι διατεθειμένοι όμως να συζητήσουν, θα συζητήσουμε κι εμείς. Δεν διαπραγματευόμαστε ε, υπό απειλή, ε, το συζητήσαμε κι αυτό, δεν διαπραγματευόμαστε εκβιαστικά, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε σημεία που ανησυχούν και τι δύο πλευρέ. Και υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε τι επόμενε ημέρε και εβδομάδε και θα επανέλθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα συζητήσω αυτά. Για τον ΠΟΕΜ. Πρέπει να λύσουμε το θέμα του ε, σώματος ε, υποβολή εφέσεων και δεν έχουμε δει καμία κίνηση από την Αμερικανική πλευρά. Κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί φυσικά αυτό απειλεί το όλο σύστημα. Δεν έχω λύση να σας προσφέρω σήμερα, αλλά ε, πρέπει να βρούμε. Επίσης πρέπει να δούμε διάφορα στοιχεία. Υπάρχει μια πολυμερής πλευρά που μπορούμε να δούμε ίσως τα θέματα αλληλείας σε πολυμερές επίπεδο ε, αποτύχαμε στον Buenos Aires, αλλά να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα. Ε, ίσως λοιπόν να κάνουμε μια πολυμερή προσπάθεια γι' αυτό. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε ένα πιο ευέλικτο ε, τρόπο πολυμερής, πολυμερούς προσέγγισης. Οι χώρες που θέλουν να συμμετέχουν με πλήρη διαφάνεια, πλήρη σεβασμό των κανόνων του ΠΟΕ και να μπορεί να συμμετέχει όποιο επιθυμεί, να λάβουμε κάποια βήματα ας πούμε. Για παράδειγμα, για το ηλεκτρονικό εμπόριο, πάνω από 70 χώρες, φτωχές και πλούσιες ε, στο βορρά και στο νότο προσυπέγραψαν και θέλουν να προχωρήσουν. σω θα μπορούσαμε να εξετάσουμε πώ να προχωρήσουμε και ίσω αυτό είναι ένα τρόπο να δούμε ε, αν ε, υπάρχει και διάθεση για τη διαδικασία. Είχατε και δύο ακόμα πιο φιλοσοφικέ ερωτήσει, θα έλεγα που είπατε αν υπάρχουν πολλές απαιτήσει στο κεφάλαιο του εμπορίου και της βιώσιμη ανάπτυξη. Πάντα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος και ορισμένες φορές με ρωτάτε γιατί δεν θίξαμε το τάδε το δίνα. Όλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά μια εμπορική συμφωνία δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου και νομίζω ότι υπάρχει παγκόσμια συνειδητοποίηση ότι οι διεθνείς συμβάσεις ε, όπως εγκρίθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη, η Συμφωνία του Κλίματος των Παρισίων, ε, τα διεθνή πρότυπα πρέπει να υπάρχουν και από εκεί και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο με κάποιες χώρες. Για παράδειγμα διαπραγματευόμαστε με το Μεξικό ένα κεφάλαιο για τη διαφθορά. Αυτό είναι καλό και ριζοσπαστικό, αλλά θα πρέπει να πιέσουμε ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες στο ευρύτερο ε, θέμα των 27 κριτηρίων που έχουν προσυπογράψει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντα όμως πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Να υπάρχει κάτι βασικό, ένα βασικό σύνολο θεμάτων με όλες τις χώρες και μετά υπάρχουν και άλλες χώρες να συνεργαστούμε και με κάποιες, και άλλους τρόπους μάλλον να συνεργαστούμε μεμονωμένα με κάποιες χώρες. Υπάρχει όμως παγκοσμίω η συνειδητοποίηση ότι το εμπόριο έχει μια πολύ ισχυρή βάση αξιών και και εμείς και άλλες χώρες το πιέζουμε. Όσον αφορά το πολυμερές δικαστήριο, υπάρχει η εντολή του Συμβουλίου. Ίσως κυρία Χάουτελα όντω δεν ήμασταν ε, αρκετά συγκεκριμένοι, είναι αρκετά δύναμο, αλλά είναι ένας τρόπος να ξεκινήσουμε. Δεν επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σύστημα με τους, στους υπολείπους, αλλά ξεκινούμε με κάποιες χώρες ανά τον κόσμο. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια κρίσιμη μάζα χωρών για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε είχαμε μια διαδικασία που είναι χρήσιμη γιατί συζητιέται το θέμα και γίνεται σε βάση Ηνωμένων Εθνών με πολλέ χώρε εκεί. Δεν σημαίνει ότι θα είναι όλε εκεί, αλλά είναι ένα τρόπο να το προωθήσουμε. Τώρα που υπάρχει εντολή, η οποία είναι η βασική εντολή με τα ουσιώδη, αλλά μπορούμε από αυτά να ξεκινήσουμε να προσεγγίσουμε χώρε και να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Και εδώ φυσικά θα εκτιμούσα και τη δική σα ε, συμβολή, αλλά και των υπολείπων. Κυρία Ρενά, ρωτήσατε για τις ε, συμφωνίες τι γίνεται. Αν δεν συμβεί τίποτα θα τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα από απόψε. Ε, περιμένουμε ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ ότι κάποιε χώρε θα εξαιρεθούν και ελπίζουμε να είμαστε στον κατάλογο. Αλλιώ ξεκινάει η σχέση του από απόψε. Και φυσικά είμαστε πάντα διατεθειμένοι να συζητήσουμε με του Αμερικανού ε, ε, εταίρου, αλλά δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα υποπίεση ή απειλή. Για τον Καναδά έγιναν κάποιε συνεδριάσει για το κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Ένα θέμα που συζητήσαμε είναι η Συμφωνία του Κλίματος για το Παρίσι. Πώς μπορούμε να το συμπεριλάβουμε και αυτό. Και νομίζω η ομάδα εργασία προβλέπει μια ακόμα συνεδρία στο Μάιο. Ίσως λοιπόν θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε μετά από αυτό. Για το θέμα του Μαρόκου. Η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση είναι αρμόδια για αυτέ τι συζητήσει. Ε, γνωρίζουμε τι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση το συντομότερο δυνατόν βεβαίω, διότι όπω είπατε ε, μα πιέζει ο χρόνο. Ε, από ό,τι ακούω οι συζητήσει βαίνουν καλώ, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Για τη Μερκοσούρ, αρκετοί ρωτήσατε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευαισθησίε στον τομέα τη γεωργίας δεν απελευθερώνεται όλο το μέσο της γεωργίας. Ε, θα ε, δουλέψουμε με ποσοστό όπως γνωρίζετε και ξέρουμε ότι υπάρχουν ευαισθησίε και κόκκινες γραμμές σε κάποιες χώρες ε, που με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά, αλλά έχουμε και επιθετικά συμφέροντα στη Μερκοσούρ και στη Γεωργία και στον Νίνο, στα γαλακτοκομικά, και σε άλλα ποτά, με ποιημένα τρόφιμα, σοκολάτα κλπ. Υπάρχουν λοιπόν και επιθετικά συμφέροντα εκεί και φυσικά ε, το ενδεχόμενο πρόσβασης σε μια αγορά 200 εκατομμύριων, 260 εκατομμυρίων ανθρώπων σε υπηρεσίες, σε δημόσιες προμήθειες κλπ. είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ευρύτερη η συμφωνία που θα κάνουμε. Οκταπλάσια της συμφωνίας με τον Καναδά, αν δείτε τους δασμούς. Για τη συμφωνία με την Ιαπωνία, Υπάρχουν διατάξει ε, για την καταπολέμηση τη παράνομη υλοτομίας που περιλαμβάνονται στη συμφωνία με την Ιαπωνία και θα τα προχωρήσουμε. Κύριε Μακλάκη, συμφωνώ μαζί σας ότι όταν συζητούμε για βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρχει μια βάση στι πολυμερεί συμφωνίε, στις διεθνεί συμβάσεις ε, των ΗΕ, συμβάσει του Διεθνού Γραφείου εργασία, Μπορεί να είναι και στοιχεία επιπλέον. Με το Μεξικό, για παράδειγμα, έχουμε το κεφάλαιο για τη διαφθορά ή και άλλα πράγματα. Μπορούν να αποτελούν όμω και μια βάση η οποία θα είναι το μοντέλο για να μπορούμε να προβλέπουμε και κάποια ε, ε, πράγματα. Αλλά με κάθε χώρα μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, συγκεκριμένα θέματα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, που να πηγαίνουν πέραν αυτών των βασικών στοιχείων. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να βασίζονται στι πολυμερεί συμφωνίε και να υπάρχει διαφάνεια σε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί την Ταϊβάν και το Χονγκ ναι, πράγματι πρέπει να υπάρχουν ε, Διαπραγματεύσει για τι επενδύσει ε, με αυτέ τι δύο χώρε και μάλιστα έχουμε προτείνει να γίνουν από κοινού. Δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ε, υπήρχε μια ομάδα εργασία και με τι δύο χώρε για να δούμε πού βρισκόμαστε. Πήγε πολύ καλά. Δεν έχουν ξεκινήσει η διαδικασία για να δούμε τι πεδίο εφαρμογή θα έχουμε. Ελπίζω να ξεκινήσει σύντομα. Για το Βιετνάμ. Κυρίως επικεντρωθήκαμε στην Ιαπωνία για τις μεταφράσεις. Οι μεταφραστικές υπηρεσίες πιέζονται πάρα πολύ, αλλά ελπίζουμε να μπορέσουν να υποβάλουν την απόφαση για την Ιαπωνία πριν από το καλοκαίρι, να την έχετε εσείς ε, πριν από το φθινόπωρο, για να την έχετε πριν από το τέλος της θητείας σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, πότε θα έχουμε την εντολή. Αυτό είναι θέμα του Συμβουλίου. Ελπίζω να απαντήσουν σύντομα, γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις πριν από το καλοκαίρι και το ελπίζουμε. Ακούω ότι πάει καλά. Αλλά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Ίσως θα μπορέσετε να το θέσετε στην Προεδρία αυτό. Κυρία Σάκχε, εμείς, ε, αν κατάλαβα καλά, τι ρωτάτε, έχουμε διευκρινίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία, θέλουμε μεταχείριση ως ένας, δεν δεχόμαστε ξεχωριστές εξαιρέσεις. Και δεν είναι πολύ εύκολο να εξηγήσουμε πάντα πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να του κάνουμε λίγο μάθημα των Αμερικανών σε διάφορα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω είναι μία, έχουμε μία εμπορική πολιτική και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα διαβιβάστηκε και όλα τα κράτη-μέλη έχουν υπάρξει ιδιαίτερα σαφή. Η ενότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονιστεί εδώ. Τώρα, θα προσφύγουμε στον ΠΟΕ. Νομίζω θα πρέπει να είναι σαφέ ότι ε, υπάρχουν όλα τα στοιχεία να προσφύγουμε στον ΠΟΕ είτε μόνοι μα είτε με για τα μέτρα διασφάλισης, διότι ε, ο κλάδος μας ούτως ή άλλως έχει πληγεί από τις διάφορες ε, παρεκκλήσεις του εμπορίου και ε, προετοιμάζουμε την ένσταση, πρέπει να την προετοιμάσουμε. Υπάρχει προθεσμία 90 ημερών προετοιμασίας, διαβούλευσης, κοινοποίησης και μετά από 90 μέρες που θα είναι έτοιμη θα δούμε αν θα τη χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει αυτό και αυτή φαίνεται να είναι και η θέση του Συμβουλίου. Δεν είναι... Ε, εκδίκηση αυτό, είναι ε, εξισορρόπηση κύριε Ντάρτμουθ και αυτό έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τον κατάλογο, αλλά πρέπει να υπάρχει στην περίπτωση που μας επιβληθούν για παράδειγμα δασμοί, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα εξαιρεθούμε, να καταρτιστεί ο κατάλογος και να δούμε αν θα το χρησιμοποιήσουμε ή όχι, ε, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η απόφαση για το ενδοκινοτικό σύστημα επίλυσης διαφορών, κυρία Χάουταλα, να σας πω ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτά ε, συνάδουμε το εσωτερικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, εσωτερικό σύστημα επίλυσης διαφορών και χαίρομαι που το δικαστήριο είπε το ίδιο πράγμα. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει επιρροή για άλλα τα δικαστηρία. Νομίζω ότι αναφέρεστε στο βελγικό ε, ε δικαστήριο για τη ΣΥΤΑ. Δεν ξέρω πότε θα το έχουμε, κατά πάσα πιθανότητα αρχέ του επομένου έτου, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου και θεωρούμε ότι είναι τελείω διαφορετική διαδικασία. Δεν υπάρχουν παρεμβολές. Για το Φινικέλο υπάρχουν ε, ε, ανησυχίες και το λέμε στου Μαλισιανού και Ινδονησίου εταίρου, αλλά έκαναν προσπάθειες για να γίνει βιώσιμη η διαδικασία. Ε, υποστηρίζουμε αυτέ τι πρωτοβουλίε, έχουμε συνεργαστεί και μαζί του σε κάποια από αυτά, έχουν στόχο να είναι πλήρως ε, βιώσιμα το 2020, κυρίω στην Ινδονησία και πρέπει να του στηρίξουμε, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά προϊόντα για αυτού και πρέπει να στηρίξουμε τη δουλειά του για να είναι βιώσιμη η παραγωγή. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα, και έχουμε ένα πολύ ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο. Του συνάντησαν πριν από κάποιες εβδομάδες και τη Μαλισσία και την Ινδονησία και το συζητήσαμε. Κύριε Σόλτς, για τις, ε, τους αποκλεισμούς εταιριών και προϊόντων υπάρχει μια τελείως διαφορετική διαδικασία που διαχειρίζονται οι εταιρείε σύμφωνα με κάποια κριτήρια. Δεν υπάρχει καμία πολιτική παρέμβαση. Ε, πάνε παράλληλα αυτά για την υπερβολική παραγωγή. Όπως είπα, εργαζόμαστε ήδη στον ΟΣΑ, στο φόρουμ του Χάλιβα, όπου καταφέραμε να συμφωνήσουμε με τους Κινέζους εταίρους μας για περισσότερη διαφάνεια και το τι κάνουν σε σχέση με αυτό. Περισσότερη διαφάνεια στις ε, κινέζικες επιδοτήσεις. Ελπίζουμε λοιπόν τον Μάιο ή τον Ιούνιο να έχουμε μια νέα συνάντηση και συμφωνήσαμε με την Ιαπωνία να συνεργαστούμε για επιβολή των κανόνων του ΠΟΕ, να δούμε αν υπάρχουν κανόνες, γιατί ο ε, ΠΟΕ δεν είναι φτιαγμένο για το είδος της οικονομίας που έχει η Κίνα και ίσως υπάρχουν και άλλες ε, περιπτώσεις ε, που μπορούμε να δούμε στο πλαίσιο της συνεργασίας και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό. IPR ναι, είναι η πνευματική ιδιοκτησία ε, ζήτημα πολύ ευαίσθητο στην Mercosur και πρέπει να το δούμε. Ε, δεν το έχουμε επιλύσει, πρέπει να βρεθεί μια λύση για την Κίνα. Έχουμε, όπως ξέρετε, διαπραγματεύσεις για τις επενδύσεις. Είναι αργές αλλά σημαντικές. Ο στόχος είναι να επιτύχουμε ένα καλύτερο καλύτερου όρου, ίσου όρου ανταγωνισμού, γιατί ε, γίνεται δυσκολότερο για τι εταιρείε μα να δράσουν στην κινέζικη αγορά. Αυτό πρέπει να το δούμε και οι επενδύσεις για τις διαπραγματεύσει είναι το φόρουμ που έχουμε. Υπάρχει κάποια πρόοδος, ε, σιγά σιγά όμως, αλλά εκεί πέρα είμαστε σε επαφή και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτές τις ε, συζητήσεις. Ε, έχουμε και την Σύνοδο Κορυφής με την Κίνα το καλοκαίρι και θα τεθούν αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω πως απάντησα στην ερώτησή σας ε, κύριε Ντόφμαν επιζητούμε εξαιρέσεις και διάλογο με τις ΗΠΑ δεν θέλουμε αντίπεινα η κλιμάκωση αλλά σε συμφωνία με το Συμβούλιο έχουμε έτοιμα αυτά τα εργαλεία αν τα χρειαστούμε. Ε, ε, μου επιτρέπετε να επανέλθω στην ερώτηση της Μαρίτιες Χάκε. Αν ε, θα πάτε σε αντίπεινα, ακόμα και αν επιτύχει εξαίρεση η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον, θα είναι κοινή αυτή η προσέγγιση με άλλους εταίρους. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει, ελπίζω απόψε, αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Αν υπάρξει πλήρης εξαίρεση. Ήμουν σε επαφή με πολλές χώρες τις τελευταίες εβδομάδες να δούμε αν θα μπορέσουμε να συντονιστούμε. Θέλουν όλοι να αναλάβουμε κοινή δράση, αλλά περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Τα, τα, Χριστού... τα... μεσάνυχτα, με συγχωρείτε, θα δούμε το τι θα γίνει. Θα δούμε λοιπόν αν θα προκύψει κάτι άλλο. Ας περιμένουμε και θα το αξιολογήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Ε, δύο λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Κέλλη πρώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Να σας συγχαρώ που φοράτε και πράσινα σήμερα είναι η εβδομάδα του Αγίου Πατρικίου στην Ιρλανδία. Να σας συγχαρώ και για τις ε, προσπάθειές σας που κάνατε στην ε, θητεία σας ως Επιτροπός ε, Εμπορίου. Έτσι ακριβώς συνέβη το θέμα με, το, με την TTIP και τελικά καταλήξαμε σε συμφωνίες με άλλες περιοχές του κόσμου. Θα ήθελα να επικεντρωθώ εγώ σε ένα θέμα, αναφέρατε την Ιαπωνία, κάτι το οποίο είναι θετικό. Θα θυμάστε όμως πριν από λίγους μήνες συζητούσαμε την ε, Σιγκαπούρη και κάποιοι συνάδελφοι ανέφεραν ότι η κατάσταση πλέον ε, γινόταν δύσκολη και μας έφερνε σε αμηχανία γιατί περιμέναμε πέντε χρόνια για μια κύρωση, είχε πάει στο δικαστήριο, η υπόθεση στο ΔΕΚ μαζί με την ΣΥΤΑ. Τώρα όμως έχει καθαρίσει και θα ήθελα να γνωρίζω εάν του δίνεται προτεραιότητα για να ολοκληρωθεί φέτος. Κάποιοι ευρωβουλευτές ήμασταν στη Σιγκαπούρη πριν από λίγες εβδομάδες ε, και για να πω την αλήθεια ήταν πολύ υπομονετική με κατανόηση αλλά θα ήθελα να πω το να τιμωρείται η Σιγκαπούρη επειδή κάποιες άλλες μεγαλύτερες ε, χώρες ε, ε, εμφανίστηκαν δεν είναι σωστό. Σας ευχαριστώ κύριο Σκάριμ. Επίτροπε. Επίτροπε, παρά το σκληρό σας πρόγραμμα ήρθατε σήμερα εδώ και αυτό δίνει, δείχνει τη σχέση σας με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας και σας ευχαριστούμε. Είμαι επικεφαλής της υποομάδας ε, για το εμπόριο με την Νότια Ασία. Θέλω να αφαιρθώ σε δύο χώρες. Πρώτα απ' όλα, πριν από λίγους μήνες, ο πρόεδρος Τούσκ πήγε στην Ινδία για να αναβιώσει την Συμφωνία Ελευθερίου Εμπορίου. Ε, έκτοτε βεβαίως σιωπή. Ε, και αυτό με ανησυχεί, γιατί είτε ε, δεν συμβαίνει τίποτα, είτε συμβαίνει κάτι και δεν το ξέρω εγώ. Και το ότι και εσείς δεν είπατε κάτι σήμερα με κάνει να σας κάνω την ερώτηση. Το ταχυδρομείο μου δέχεται πάρα πολλές ερωτήσεις για το τι γίνεται στο Κασμίρ αυτή τη στιγμή όπου χρησιμοποιούνται πλαστικές σφαίρες που τυφλώνουν και τραυματίζουν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας λένε το τι γίνεται, αλλά δεν έχουν πρόσβαση, οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία ενημέρωση για τις συνομιλίες. Δεύτερον, σε σχέση με τον Μπαγκλαντές, δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα το Μπαγκλαντές ε, έχει το θέμα των προσφύγων Ροχίνγκια. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να έχει κάποιο μεγαλύτερο περιθώριο στα εμπορικά για να τους βοηθήσουμε με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πέρα από τη βοήθεια που δίνουμε. Και η κυβέρνηση εκεί θέλει να πάει από το καθεστώς ε, ελάχιστα ανεπτυγμένων χωρών στις χώρες μέσου εισοδήματος. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε ε, να τους βοηθήσουμε να περάσουν και στο καθεστώς ε, γενικευμένων προτιμήσεων. Είχα πάει πρόσφατα στο Μαγκλαντές. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεργαζόμαστε μαζί τους για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Μπουχνέρ. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω, ευχαριστήσω που είσαστε εδώ πέρα και που αφιερώνετε το χρόνο σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτη ερώτηση. Τι γίνεται με τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Έγινε το περιστατικό στη Φουκουσίμα και πριν από δύο χρόνια αποφασίσαμε μέσω κανονισμού ότι οι αξίες ε, ακτινοβολίας είναι όπως τις έχουμε προεισδορήσει σε περίπτωση ε, πυρηνικού συμβάντος. Θέλω να ρωτήσω, ε, χρησιμοποιούμε αυτόν τον κανονισμό ε, για τη μελλοντική συμφωνία με την Ιαπωνία. Από επίσημα στοιχεία της γερμανικής κυβέρνησης έμαθα ότι ε, αν χρησιμοποιούσαμε αυτό τον ε, κανονισμό σε περίπτωση Ευρωπαϊκού Πυρηνικού Συμβάντος θα είχαμε 900 νεκρούς ε, παραπάνω. Δεύτερη ερώτηση. Τι γίνεται με την εφαρμοσιμότητα των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος στις οποίες αναφερθήκατε. Ε, σε σχέση με τη Συμφωνία του Παρισιού, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν ε, κάποιες ε, νομικές ε, δυνατότητες να εφαρμόσουμε αυτές τις διατάξεις και σε σχέση με την συμφωνία με το Μερκοσούρ είναι ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα. Παραδείγματο χαρή αποψηλώνεται ε, με πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του τροπικού δάσους ε, για την καλλιέργεια της ε, σόγια, κυρίως για να εξαχθεί στην Ευρώπη. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Υπουργός Γεωργίας της Βραζιλίας είναι κάτοχος μιας δασικής έκθεσης που είναι μεγαλύτερη από την Ισπανία. Ε, τρίτη ερώτηση. Τι γίνεται σε, ως προς την νομοθετική συνεργασία και με την Ιαπωνία όπως σας είπα αλλά ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, συμφωνία του Mercosur Regulatory Cooperation ε, ρυθμιστική συνεργασία. Τι γίνεται στη, στη, σχέση μας με το Mercosur. Ευχαριστούμε. Δεν καταλάβατε την πρώτη ερώτηση. Καταλάβατε. Ωραία. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο για την παρουσία της. Να σας συγχαρώ και εγώ για την ε, προσπάθεια που κάνετε για να ε, δείτε το θέμα των σχέσεων ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή αναφέρθηκαν τα περισσότερα θέματα, θα ήθελα να σε κάτι άλλο. Έχω ένα εμπιστευτικό έγγραφο, αλλά όπως θα γνωρίζετε από την εκστρατεία Stop Ψέτα, δημοσιοποιήθηκε για την ε, συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών που θα γίνει 26 Μαρτίου στον Καναδά. Είναι μία από τις πολλές συνεδριάσεις και κλεισμένο των θυρών που προβλέπονται από τη ΣΕΤΑ, αλλά σε αυτή τη συνάντηση θα συζητηθούν και τα φυτοφάρμακα επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια μας ε, διαβεβαίει ότι είναι ε, ανώδυνες ανταλλαγές απόψεων αυτές τις συναντήσεις, αλλά βλέπουμε το Καναδάς από την πρώτη μέρα ζητά να συζητήσουμε περιορισμούς για τις χημικές ουσίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείται η γλυφοσάτη σε, πολλά ευρωπαϊκά χρόνια, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και τη χρήση ενός επικίνδυνου άλλου φυτοφαρμάκου. Και πραγματικά εγώ νομίζω, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς κυρία Επίτροπε, είναι μια ομάδα ποιησης. Έχουμε εκπροσώπους του κλάδου, αλλά δεν έχουμε ρετούς ε, ε, βουλευτές ε, που να συμμετέχουν σε αυτή τη συνεδρία και να διασφαλίσουν το δημοκρατικό έλεγχο. Ε, ξέρω την άποψή σας ότι αυτά δεν είναι νομοθετικά όργανα και συμφωνώ αυτές τι συναντήσεις, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι εγώ δεν νιώθω άνατα με συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών που συζητούνται πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε ή να μειώσουμε και να διαγράψουμε πρότυπα τα οποία είναι προς όφελος της υγείας μας. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σα για το θέμα και κυρίως πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια σε αυτές τις συναντήσεις. Ευχαριστώ. Πέντρο Σίλβα, ευχαριστώ. Ε, δύο ερωτήσεις, μία λεπτό ε, ένα λεπτό ερώτηση για τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ. Φυσικά, φυσικά υποστηρίζουμε την Επίτροπο, όχι μόνο εμεί οι σοσιαλιστέ, αλλά πιστεύω ότι ε, σύσσωμο το κοινοβούλιο, τουλάχιστον η πλειοψηφία του, θα πρέπει να περιμένουμε την εξαγγελία τη κυβέρνηση. Όμω θέλω να αναφερθώ σε αυτά τα συγκεκριμένα αιτήματα που υπέβαλε ο Πρόεδρο Τραμπ για να χορηγήσει την εξαίρεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτού, αυτά τα δοσμολογικά μέτρα. Θέλω να ξέρω εσείς πώς ανταποκριθήκατε σε αυτά τα αιτήματα. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΣΥΠΑ ΕΕ που θα κρύβεται ε, πίσω από αυτή την εξαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα προστατευτικά δοσμολογικά μέτρα δεύτερον. Επειδή είμαι ο ε, μόνιμος ε, για την ε, συμφωνία με την Ιαπωνία και επειδή αναφερθήκατε σε αυτή θέλω να ρωτήσω εάν ε, προβλέπει τη ημερομηνία για την υπογραφή της συμφωνίας αναφέρθηκε ο Ιούλιος μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτή τη, αυτό το χρονικό ορίζοντα και για το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε αυτή τη συμφωνία θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξήγηλε 15 δράσεις για να καταστούν αποτελεσματικότερα τα κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, προβλέπεται ήδη ε, αυτό το κεφάλαιο να συμπεριληφθεί και στο συμφου... στη συμφωνία με την ε, Ιαπωνία. Και ποια η σχέση με την κοινωνία των πολιτών και τι θα γίνει με τη ρήτρα αναθεώρησης που θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Ευχαριστώ, Γιώχη Σούστερ. Ευχαριστώ. Ε, τους ε, τελευταίους μήνες κάναμε συζήτηση για ε, την εφαρμοσιμότητα του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι πρέπει να γίνεται, ότι δεν υπερασπίζεται αυτή την αξιολόγηση, δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια Έχουν φυλακιστεί ε, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, ε, οπότε για την εφαρμοσιμότητα αυτών των κεφαλαίων βιώσιμη ανάπτυξη αναρωτιέμαι εγώ. Ε, τι επόμενε εβδομάδε τον τελευταίο μήνα, ε, θα ενεργοποιήσετε αυτό το μηχανισμό διευθέτησης ε, διαφορών μέσα στο κεφάλαιο ή πώς ε, προβλέπετε εσείς να εφαρμόσετε αυτό το κεφάλαιο. Ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Πώς σκοπεύετε να εξασφαλίσετε την εφαρμοσιμότητα αυτού του κεφαλαίου. Είναι θέμα αξιοπιστίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή τον είτε στα σοβαρά ή πέρα από τα μεγαλόσχημα λόγια δεν συμβαίνουν και πολλά πράγματα τελικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον Επίτροπο που ήρθε στην Επιτροπή μας ε, για τις ε, προσπάθειες που καταβάλλετε για τις συμφωνίες ελευθερίου εμπορίου. Ξέρω πως έχουμε ζητήματα με τις ΣΥΠΑ, με την Κίνα και τις μελλοντικές εμπορικές ε, συμφωνίες. Τώρα όμως έχουμε αυτόν τον δομημένο διάλογο και μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Έχω κάποια σχόλια για τις σχέσεις μας με την Νορβηγία και τις επιπλέον ε, εμπορικές ε, προτιμήσεις στα γεωργικά προϊόντα. Το πρωί το ψηφίσαμε αυτό και αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι πως η Νορβηγία μετά από τις ε, διαπραγματεύσεις μας επέβαλε νέους δασμούς ε, στα λουλούδια και παρά το ότι εμείς ε, δεσμευτήκαμε όπως και η Νορβηγία στην περαιτέρω απελευθέρωση θεωρώ ότι στην συζήτηση που κάναμε στις 20 Φεβρουαρίου και με τον Νόρβηγο πρέσβη, τον ρωτήσαμε γιατί το έκανε αυτό και μας είπε είναι τεχνικά αυτά τα ζητήματα, μας υποσχέθηκε όμως ότι θα έστελνε μια επιστολή προς την Επιτροπή, την οποία δεν λάβαμε και νομίζω ότι η Νορβηγία ξεκάθαρα διαπραγματεύεται κακόβουλα το είδαμε το 2010 όταν ε, ξαφνικά μία ημέρα είχαμε δασμούς ε, σε βόηο χοιρινό κρέας ε, και λουλούδια. Αντιλαμβάνομαι πως είχαν γίνει αυτές οι συμφωνίες και από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αλλά πρέπει να συντονίζονται οι υπηρεσίες σας. Υποτίθεται ότι είμαστε μεγάλο εμπορικό μπλοκ. Αν μπορούν δηλαδή να μας ε, ξεγελάνε και οι μικροί εταίροι γιατί οι διάφορες γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν δεν συντονίζονται, δεν ξέρω τι γίνεται. Ελπίζω να επιληφθείτε του θέματος και να έχουμε κάποια απάντηση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά. Ε, επιμένετε σε αυτό το θέμα. κύριος Σταρμπάτη. Σεβασμό, τον σεβασμό μου να εκφράσω κύριε Επίτροπε που παρακολουθείτε όλα τα θέματα. Ε, έχω κάποιες ε, ερωτήσεις. Ε, εντάξει, ελπίζουμε να υπάρξει κάποια εξαίρεση, αλλά αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ είναι και θέμα αρχής. Ε, λένε οι οικονομολόγοι ότι πρόκειται για προστατευτισμό, για να προστατεύσει την οικονομία του, οπότε θα επανέλθει αυτό και αναρωτιέμαι εάν η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει πρωτοβουλία και να πει εάν θέλει να αποκλείσει τη χώρα του ο Τραμπ, εμείς θα ανοίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στον κόσμο. Να πούμε, ας πούμε, ότι θα μειώσουμε τους δασμούς μας α, ε, ε, για τα αμερικανικά αυτοκίνητα που είναι 10% ε, οι δασμοί, ενώ η δική μας προς τη ΣΥΠΑ είναι 2% αυτό πραγματικά θα ήταν μια όθηση κατά του κυρίου Τραμπ και όθηση του ελευθέρου εμπορίου. Μία ερώτηση κάτω μου προς την κυρία Ρόβολτ. Αντιλαμβάνομαι ε, αυτά τα οποία λέτε φιλοσοφικά ότι δεν μπορούμε να βάλουμε όλες μας τις ευρωπαϊκές αξίες, τις εμπορικές συμφωνίες. Γνωρίζουμε από εμπειρία πως οι αξίες και οι θεσμοί είναι θέμα ιστορικών εξελίξεων. Έχει προχωρήσει η Ευρώπη και δεν μπορούμε να περιμένουμε όλος ο κόσμος να ακούει τις ευρωπαϊκές εντολές. Αλλά άκουσα και εδώ πέρα κάποια πράγματα που α, σκεφτόμουν να μοιάζει αυτό λίγο με ευρωπαϊκό υπεριαλισμό να τα κολλάμε όλα αυτά στο εμπόριο. Ε, όχι, εντάξει, και οι μπεριαλιστές. Ραμόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση έχω μόνο. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά σας ε, και εμείς ως φιλελεύθεροι είμαστε υπερήφανοι για το πώς αντιμετωπίζετε τα διάφορα θέματα. Ταξιδεύετε ανά τον κόσμο, δεν είναι εύκολο. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε. Μία ερώτηση για την Σιγκαπούρη. Πήγατε εκεί πριν από λίγες εβδομάδες ε, και οι βουλευτέ είχαν πάει πριν πάτε εσεί. Μπορούμε να περιμένουμε κάποιο κείμενο το καλοκαίρι γιατί ε, από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσουμε. Η Συμφωνία Εμπορίου περιμένει από το 2014. Ε, έχουν απογοητευτεί στην Σιγκαπούρη. Χάνουμε χρόνο. Και νομίζω ότι είναι υποφελέ για όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε γιατί δεν εξάγουν τίποτα σε εμά, δεν παράγουν αυτοκίνητα, ούτε γεωργικά προϊόντα. Είναι υποφελές λοιπόν. Πώς α, μπορούμε να περιμένουμε θετικά νέα σε αυτό το μέτωπο και είμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και να συμφωνήσω κι εγώ με όλου του συναδέλφου και να σα συγχαρώ γιατί ήρθατε απευθεία μετά από το ταξίδι στα στην και να σα συγχαρώ και για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε διότι από την αρχή αυτή τη θητεία μέχρι τώρα έχει γίνει πολλή ε, δουλειά, έχετε κάνει πολύ μακρύ δρόμο, μας μένει κι άλλους ακόμα αλλά έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Όσον αφορά το ε, εμπόριο για την ανάπτυξη, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι δύο κανονισμοί που εγκρίθηκαν και για τα ορυκτά σε περιοχές ε, σύγκρουσης αλλά και για τα θέματα της θανατικής ποινής ε, ε, και είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την πολυμερή διάσταση αλλά ήθελα να ρωτήσω μήπως θα έπρεπε στις διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες να συμπεριληφθεί και η δέσμευση να γίνει αποδεκτός αυτοκανονισμός και για τα ορυκτά σύγκρουσης και για το εμπόριο για να μην εμπορεύονται Υπάρχουν εργαλεία για βασανισμούς και θανατική ποινή. Και επίσης ε, θα μπορούσε να είναι καταρχάς μια δέσμευση από πλευρά τους ε, το να συμπεριληφθούν αυτά ε, στις συμφωνίες. Τώρα, όσον αφορά την Ιαπωνία, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε ίσως ένα κεφάλαιο ή μάλλον μια συμφωνία για τις επενδύσεις διότι νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία με την Ιαπωνία σε θέματα επενδύσεων και ε, αν υπάρχει δυνατότητα πώς θα μπορούσε να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Τώρα όσον αφορά την κατάσταση στις Ηνωμένε Πολιτείες νομίζω ότι ήταν σαφές ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, δεν είχαν θεωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αυτό που είναι εταίρος σύμμαχος και νομίζω ότι δεν υπήρχε κίνηση ε, για την εθνική ασφάλεια, αλλά για πολιτικούς λόγους από πλευράς Τραμπ, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με θέματα εμπορίου αυτά που κάνει. Και επίσης ε, ελπίζω να ανακοινωθεί ε, κάτι θετικό για μας, όπως ελπίζουμε όλοι, και η ερώτησή μου είναι εξής το να ανταποκρίνεται σε κάποια θέματα για πολιτικούς λόγους θα μπορούσε να πλήξει και άλλους τομείς. Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει σε θέματα δασμός, ε, δασμών ο κύριος Τραμπ, ο κύριος Τσίκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνει και κυρίως να τονίσουμε και ότι η Ευρώπη ενωμένη μπορεί να ε, σταθεί ε, απέναντι σε αυτούς του τύπου τις ανταπαραθέσεις. Και να πω ότι, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ότι όσον αφορά την απόφαση του Τραμπ απόψε, θα υπάρχουν και άμεσες συνέπειες ε, και έμεσες συνέπειες. Οι άμεσες συνέπειες είναι ό,τι αφορά την επιβολή δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όπως και να έχει, ε, υπάρχει το μεγάλο θέμα και το μεγάλο πρόβλημα των έμεσων συνεπειών, διότι θα υπάρχει ένας επαναπροσανατολισμός σε εμπορικό επίπεδο με το χάλιβα. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Τουρκία σήμερα εξάγει στις ε, αμερικανικές αγορές πάνω από 200.000 τόνους, 200 ε, τόνους ε, χάλιβα. Αν κλείσει η αμερικανική αγορά, αυτές οι 200.000 τόνοι θα στραφούν προς την ευρωπαϊκή αγορά. Και ναι, μεν αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να περιμένουμε, να δούμε προσεκτικά τι κινήσεις θα κάνουν οι υπόλοιποι, αλλά υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι βέβαιες και προβλέψιμε. Και δεδομένες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε δώσει κάποιες απαντήσεις από τώρα ε, πέραν της διαδικασίας των 90 ημέρ και ε, των 90 ημερών και πέραν της σωστής και πολύ προσεκτικής εκτίμησης που πρέπει να κάνουμε για να δούμε πώς θα προσανατολιστούν οι υπόλοιποι. Να μην μιλήσω δε για την Κίνα που ήδη από σήμερα έχει εξαγωγές διπλάσιες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Επομένως, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή την πτυχή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τα άλλα θέματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, αλλά υπάρχει σήμερα ο κλάδος μας, ο οποίος ε, λόγω αυτών των έμεσων συνοπιών μπορεί να καταρρεύσει και να έχουμε μια κρίση και αυτό να στοιχήσει χιλιάδες ε, θέσεις εργασίας και να κλείσουν επιχειρήσεις μας. Πρέπει λοιπόν να τα προφυλάξουμε όλα αυτά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Προύστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ σήμερα. Ένα θέμα το οποίο ίσως να σας εκπλήξει και δεν ε, περιμένω και μια απάντηση ουσίας, διότι ε, οι περισσότεροι θαυμάζουμε το πώς καταφέρετε να ασχοληθείτε με όλα τα θέματα, αλλά μέρα πάντα με αποσχολεί το ίδιο. Και αφορά τον τρόπο πώς θα καταφέρετε βράχη, μέσο και μακροπρόθεσμα διότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάτι συγκεκριμένο με τις υπηρεσίες σας για τις συμφωνίες ελευθέρων εμπορίου, ε, ελευθέρων συναλλαγών και να υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό κλίμα για τις, που είναι απαραίτητο για τις επιχειρήσεις μας και πώς μπορούμε να ελοπίσουμε όμως τις μελλοντικέ συμφωνίες, πώς να διαχειριστούμε τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί, διότι μια συμφωνία ναι μεν πρέπει να υπογραφεί, το πιο σημαντικό είναι να γίνεται σεβαστή. Και όταν διαπιστώνουμε τα όσα μας περιμένουν. Και μάλιστα τα όσα είπε ο μόλις ο συνάδελφος ε, Τσίκου και είδαμε τη νέα μεθοδολογία, την ομαδική ε, και πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά αυτή τη μεθοδολογία πώς ε, αύριο ή στο τέλος του έτους θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη μέθοδο screening σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα προποθέτει και εμπλοκή των δικών σας υπηρεσιών. Πιστεύετε ότι σήμερα υπάρχει κατάλληλο ε, ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσετε να απαντήσετε σε όλα τα προβλήματα και να αντιδράτε σε όλα τα μέτωπα. Ε, και αυτό πηγαίνει πέραν των ερωτήσεων του Κοινοβουλίου ναι, μεν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πολύ συχνά χρειάζεται και κατάλληλο προπολογισμό. Αλλά εμά μα ανησυχεί. Διότι όταν βλέπω τον όγκο τη δουλειά, αν πραγματικά θέλουμε να δράσουμε αποτελεσματικά, πρέπει οι υπηρεσίε σα να έχουν αρκετού υπαλλήλου και ορισμένε φορέ ε, έχουμε και το δικαίωμα να έχουμε και κάποια ερωτηματικά από αυτού. Ωραία, ευχαριστώ. Η Επίτροπος. Ε, thank you Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αρχίσω με τον κύριο Κέλλη. Ναι. Πολύ σημαντικό είναι να συνάψουμε αυτές οι και συμφωνίες ε, τώρα λόγω της συγκυρίας, γιατί κάποιοι κλείνουν τις αγορές τους, εμείς ανοίγουμε. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κύκλο φύλων με αμοιβαίως επικερδείς εμπορικέ συμφωνίες, με κεφάλαια βιώσιμης ανάπτυξης, προς όφελος των υπηκών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλος ιδιαίτερα σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε επίγνωση των προβλημάτων και των κινδύνων που υπάρχουν, όμως είναι ε, σημαντικό στοιχείο και της ευημερίας και της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Στρέφονται οι εταίροι προς εμάς για εμπορικές ε, συμφωνίες για να συνεργαστούν μαζί μας σε πολυμερή φόρα κτλ. Για την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, πολλοί ρώτησαν για αυτά. Ε, θα... Στις 17 Απριλίου θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Σιγκαπούρη και αν έχει ολοκληρωθεί και η μετάφραση για την Ιαπωνία θα αποφασίσουμε και για την Ιαπωνία. Ε, γίνονται συζητήσει ε, για μια σύνοδο με την ε, Ιαπωνία. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η ημερομηνία διεξαγωγή. Φυσικά θα το επιβεβαιώσει και το Συμβούλιο με το που το στείλουμε. Οπότε ε, πρέπει να δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστούν και εκείνοι. Θα το στείλουμε και σε εσά ε, για να αρχίσετε την, ε, έστω και ανεπίσημα την προπαρασκευαστική εργασία. Πρεσεζίν το λένε στα γαλλικά. Και μέχρι το τέλος του τρέχοντος ή αρχές του 19 νομίζω θα έχει κλείσει το θέμα ε, για την Ιαπωνία. Για την ε, Σιγκαπούρη δεν νομίζω να. Η ίδια διαδικασία μάλλον ε, δεν νομίζω να γίνει σύνοδος αλλά θα ζητηθεί η υπογραφή οπότε ταυτόχρονα σχεδόν θα τις πάρετε. Για το Βιετνάμ λίγο αργότερα γιατί ακόμη δεν έχει μεταφραστεί. αλλά ε, ε, ακολουθούμε το χρονοδιάγραμμα. Για την Ινδία κύριε Καρύμ. Τίποτα δεν ήθελα να κρύψω. Απλώς ασχολήθηκα μόνο με τα μεγαλύτερα θέματα. Ε, στη Σύνοδο οι ηγέτες ε, συμφώνησαν να διερευνήσουν τις ε, πιθανότητες γιατί κολλήσαμε την περασμένη φορά και όπως ξέρετε και δεν θέλαμε να ξαναρχίσουμε αν δεν ξέρουμε πού τοποθετούν τις φιλοδοξίες μας. Οι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων τον Νοέμβρη συναντήθηκαν και μια νέα σύσκεψη προβλέπεται για τον Απρίλιο για να γίνει απολογισμός των πεπραγμένων και για να συνεργαστούν όσο περισσότερο γίνεται ώστε να υποβάλουν αναφορά στους ηγέτες στην επόμενη σύνοδο Σύνοδο, δεν ξέρω πότε θα διεξαρθεί, αλλά νομίζω κατά τη διάρκεια του 2018. Είναι επικοδομητική η εταίρη μας από την Ινδία, ακόμη όμως δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας, ε, οπότε θα πρέπει να δούμε αν είναι εφικτό για να μην επαναλαμβάνουμε τις διαδικασίες. Πάντως σημειώνεται πρόοδος και μετά τη σύσκεψη τον Απρίλιο των επικεφαλής των διαπραγματεύσεων θα έρθω να σας υποβάλω αναφορά πεπραγμένα. Ε, για το Μπάγκλαντες, ε, το θέμα των ε, προσφύγων. Φυσικά υπάρχει επιστήριξη. Δεν έχω τα νούμερα τώρα να σας τα πω, αλλά μπορώ να σας τα στείλω. Ε, για το εμπορικό ζήτημα. Μα απασχολεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Παγκλαντέ. Το παρακολουθούμε το ζήτημα μαζί με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ε, και την DG Empli γιατί την ε, σχετίζεται και με το εργατικό δίκαιο και τα δικαιώματα. πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για το σύμφωνο έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα σχέση μας με τον Παγκλαντές αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχει πολύ ρυθμιστική συνεργασία, regulatory cooperation όπως είπατε, ε, όπως με, στην, με την Ιαπωνία και τον Καναδά, για την αποψήλωση. Ναι, γνωρίζουμε το πρόβλημα. Για να λάβει δέσμευση για την αποψήλωση ε, στο Συμφωνία του Παρισιού στα πλέντη στις, στις υποσχέσεις της η Βραζιλία στους στόχους της ε, και γίνεται μελέτη αντικτύπου ε, για το Μερκοσούρ αυτή τη στιγμή θα συζητηθεί. Μέχρι το καλοκαίρι θα κατατεθεί η πρώτη έκθεση και μετά θα ακολουθήσει η πλήρης μέχρι το τέλο του καλοκαιριού, ούτω ώστε να αρχίσουν διαβουλεύσει με την κοινωνία των πολιτών για αυτό το θέμα και θα διαβάσουμε τα αποτελέσματα. Η εισαγωγή στροφίμων τροφίμων από την Ιαπωνία 12 δήμοι έχουν πολύ αυστηρού ελέγχου για την εισαγωγή και κάθε παρτίδα έπρεπε να ε, συνοδεύεται από τη δήλωση ότι είναι ελεύθερη ε, ραδιενέργεια ε, και δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με αυτό. Κύριε Σίλβα Ντεφερέ, δεν έχουμε καμία μυστική συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ. Είπαμε. Και νομίζω του πείσαμε ότι δεν είμαστε άπειλοι για την εθνική ασφάλεια, για το αλουμίνιο και για τον χάλιβα. Έχουμε στείλει πάρα πολλά στοιχεία και ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί στις επαφές μας και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα εξαιρεθούμε. Δεν είναι συμβατά πάντως τα μέτρα με τον, τους κανονισμούς του ΠΟΕ. Και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Είπαμε ότι θα συστηθεί ομάδα εργασία. Ε, η ακριβή σύνθεση και η μερίσια διάταξη είναι θέματα υποσυζήτηση. <clears throat> Trade irritants ε, ή ε, ευρύτερα ζητήματα, έλεγχος των επενδυτών, συνεργασία για την υπερδυναμικότητα, για την Κίνα, τι μπορεί να κάνει η Κίνα κτλ. Θα τα δούμε Λεπτομερό στο μέλλον, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για και καλυμμένη συμφωνία ή δεν είναι απειλή αυτό. Είναι ομάδα εργασία. Θα δούμε υπό ποιους όρου θα εργάζεται. Δεν υπάρχει μυστική συμφωνία με του Αμερικανού. Για την Ιαπωνία πιστεύω σας είπε για το SDS είναι το κεφάλαιο μέσα στη συμφωνία. Μπορούμε να ε, ενσωματώσουμε και ενισχυμένα μέτρα. Αυτές οι 15 δράσεις εφαρμόζονται σε όλες τις συμφωνίες, ε, στις τωρινές και τις μελλοντικές. Και πιέζουμε σκληρά την ε, ε, η Ιαπωνία για τις εκκοινοποιήσεις σε διεθνείς οργάνωσης εργασίας, για την Για την Κορέα ε, συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Εμπορίου. Ε, πολλές φορές τηλεφωνικά το συζητήσαμε, το ξέρουν. Ε, έχουμε ήδη κοινοποιήσει την ανησυχία μας και αν δεν σημειωθεί πρόοδος θα ζητήσουμε να γίνουν επίσημες διαβλέψεις για το ζήτημα. Θα περιμένουμε όμω για λίγο για να Α, δούμε. Μπορεί να προγραμματίσουν κάποια δράση. Αν όχι, θα κάνουμε μια κοινοποίηση για την ανησυχητική κατάσταση. παρότι ο πρόεδρος μας έχει διαβεβαιώσει ότι θέλει να τις υπογράψει συμβάσεις Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ε, για την Ορβηγία. Κύριε Μπένσον. ναι. Ξέρω τα περί για τα λουλούδια. Το συζήτησα με τον Υπουργό ε, εδώ και καιρό, αλλά άλλαξε η κυβέρνηση. Μπορούμε να το ξαναθέσουμε το ζήτημα και σίγουρα θα έρθω σε επαφή με τους ε, αρμόδιους συναδέλφους ε, στην Επιτροπή ε, τι γίνεται. Δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω, αλλά άμα λέτε ότι δεν το έχουμε συντονίσει το ζήτημα, του ε, σημειώνω, δεν είμαι ειδική σε αυτό το τομέα. Θα το ελέγξω. Παληθεύσω με τους συναδέλφους και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σιγκαπούρη... Το απάντησα αυτό ήδη. Καρπερή για τους δασμούς. Ε, προσπαθούμε να αποφύγουμε τους δασμούς όταν δεν έχουμε ε, συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία. Είναι το Most Favored Nation. Αυτή η ρήτρα είναι η ίδια για όλους 10% οι, οι δασμοί. Ε, εκτός ε, από τις χώρες όπου έχουμε διαπραγματευτεί συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Αντίστοιχα έχουν και εκείνοι δασμούς οι Αμερικανοί, πολύ ψηλότερους σε ορισμένες περιπτώσεις, φορτηγά, ε, ημιφορτηγά, παπούτσια, ε, κλωστοϊφαντουργικά, διάφοροι δασμοί. Αν θέλετε να ε, αφαιρέσετε τους δασμούς για τα αυτοκίνητα, θα πρέπει να τους ε, απαλείψετε για, ε, σε σχέση με τις άλλες χώρες. Δεν μπορώ να σας πω <laughs> τίποτα τέτοιο και ούτε και Ούτε και νομίζω ότι οι Γερμανοί συμπατριώτε θα, θα ενθουσιάζονταν με αυτή την πρόταση, αλλά... Δεν μπορούμε, λέμε, μας πιέζουν για να ε, καταργήσουμε τους δασμούς σε δύο εβδομάδες. Δεν, δεν γίνονται αυτά. Για οποιοδήποτε άλλα στοιχεία με ρωτήσατε, νέα στοιχεία από πλευρά Τραμπ, πού να ξέρουμε. Ε, μιλήσαμε για το Χάλιβα, είναι πολύ... Είναι θέμα πηγή μεγάλη ανησυχία για τη ΣΥΠΑ. Ε, το συζητήσαμε. Τώρα, αν θα έρχονται νέε προτάσει, πού να ξέρουμε. Για τα ορυκτά από εμπόλεμε ζώνε. Δεν νομίζω ότι γίνεται να τα συμπεριλάβουμε σε εμπορικέ συμφωνίε γιατί χρειάζεται ε, πολλή παρακολούθηση, προγραμματισμό, πόροι. Δηλαδή οι ίδιες οι χώρε πρέπει να έχουν τα μέσα για να παρακολουθήσουν την κατάσταση και να ελέγξουν την εφαρμογή. υπάρχει παγκόσμια ε, συμμαχία για, τα, ε, για τέτοια προϊόντα δεν ξέρω αν μπορούν να επιβληθούν οι κυρώσει το Σεπτέμβριο είναι η επόμενη σύνοδο. Δηλαδή, ε, καλύτερη πιθανότητα έχουμε να χρησιμοποιήσουμε τι θελωνιακέ αρχέ για να μπορούν να ελέγχουν και να επιβάλλουν ε, τι ε, κυρώσει. Για τα ορυκτά από εμπόλεμε ζώνε όμω πολύ αμφιβάλλω, γιατί σα λέω χρειάζονται πολλοί πόροι. Η ε, πονία και οι επενδύσει να συνεχίζονται αυτέ οι διαπραγματεύσει ε, παράλληλα. Χρειάζεται λίγο χρόνο αλλά δεν έχουν κολλήσει, συνεχίζονται. Το δυσκολότερο θέμα είναι το δικαστήριο των επενδύσεων. Αυτό συζητάμε, αλλά σημειώνεται πρόοδος ε, και ελπίζω να καταλήξουμε κάπου. Κύριε Τσίκου, ναι, γνωρίζουμε ότι ήδη πολλή χάλιβας που θα πήγαινε στη ΣΥΠΑ ε, ή άλλος ε, χάλιβας έχει πιθανώς κατευθυνθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλες χώρες. Η διστρέβλωση της αγοράς υπάρχει. Είμαστε σε στενή επαφή με την βιομηχανία, την Eurofair και άλλους και την βιομηχανία του αλουμινίου. Τους έχω συναντήσει και θα τους ξανασυναντήσω και μας λένε ότι το βλέπουν αυτό ήδη. Οπότε ξεκινήσαμε τις έρευνες και ίσως υπάρχουν λόγοι να επιβληθούν ακριβώς οι δικλείδες ασφαλείας ανεξαρτήτως του τι γίνεται γιατί η αγορά έχει ήδη αντιδράσει. Οπότε είμαστε έτοιμοι, έχουμε ξεκινήσει έρευνες για αρκετά προϊόντα. Κύριε Προύστ, έχετε απολύτως ε, δίκιο. Διότι βεβαίως ε, δεν είναι απλώς η διαπραγμάτευση των συμφωνιών, αυτό είναι το δύσκολο, αλλά ε, με τη στήριξή σας και τη βοήθειά σας έχουμε περισσότερες δεσμεύσεις και για την εφαρμογή των κείμενων συμφωνιών. Διότι είναι πολύ καλή διαπραγμάτευση μια συμφωνία, είναι πολύ ωραία στο χαρτί, αλλά ιδιαίτερα οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα και αν δεν μπορούν, ε, τότε δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τα κράτη-μέλη, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε βήματα, ιστοσελίδε για να μπορούν να γνωρίζουν τι δυνατότητέ του και προσδίδουμε μεγαλύτερη σημασία στην εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Δημοσιεύσαμε μια έκθεση πριν από κάποιου μήνε και συνεχίζουμε να δημοσιεύουμε ε, κάθε χρόνο τις εκθέσεις ε, και έχουμε τα σχέδια, υπάρχει ο ΠΟΕ, ε, θα έχουμε και τους Βρετανούς φίλους μας ε, σε σύντομο χρόνο. Οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Trade δουλεύουν νυχθημερών, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί, πάρα πολύ αξιόλογοι, αλλά φυσικά θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερους ανθρωπίνους πόρους. Εάν το Κοινοβούλιο λοιπόν μας στηρίξει στις διαπραγματεύσεις στον προπολογισμό, Πολύ ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και βεβαίω. Βεβαίω είμαστε στο πλευρό σας όσον αφορά τους πόρους της γενικής σας Ε, Πάντα ζητάτε περισσότερα, αλλά όπως ξέρετε δεν είναι εύκολο αυτό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας δώσατε την εικόνα και που απαντήσατε στι ερωτήσει. Ε, και παρακαλώ να παραμείνετε σε επαφή και καλή τύχη στι διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ. So, if anybody... Λοιπόν, εάν ε, θέλει κάποιος να φύγει παρακαλώ, ε, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί, αλλά εάν θέλει κάποιος ε, παρακαλώ ήσυχα. Περνάμε στο σημείο 20. Οι δραστηριότητες της παρακολούθησης των ομάδων Είχαμε την ομάδα παρακολούθησης των ΙΠΑ που στις 6 Μαρτίου συζήτησε το θέμα του Κάλιβα. Ακούσαμε τώρα τις τελευταίες εξελίξεις από την Κομισιόν. Στις 7 Μαρτίου είχαμε την ομάδα παρακολούθησης της Ιαπωνίας. Πέντρο, ναι, ευχαριστώ. Ε, συναντηθήκαμε με τον Μάουρο Πέτριτσον τελευταία φορά καθώς πλέον άλλαξε θέση. Συζητήσαμε το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά κυρίως το χρονοδιάγραμμα και θα ήθελα να σας δώσω κάποιες σχετικές πληροφορίες. Να σας πω ότι μόλις ακούσαμε ότι η Κομισιόν θα εγκρίνει την πρότασή της ε, τον Απρίλιο και το Συμβούλιο αναμένεται να υπογράψει την συμφωνία πριν από το καλοκαίρι και θα έχουμε τους όρους για να ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση. Το κείμενο υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούμε. να γίνει μια δημόσια πολιτική συζήτηση για τα θέματα αυτά. Οπότε θα έχουμε τις ομάδες παρακολούθησης ε, τον Απρίλιο και τον Μάιο και αναμένουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την... στην Επιτροπή μας τον Ιούνιο και να έχουμε μία δημόσια κρόαση τον Ιούλιο. Σκοπεύω να παρουσιάσω ένα σχέδιο σύστασης και το σχετικό ψήφισμα αμέσως ε, μόλις έρθει η συμφωνία στο Κοινοβούλιο για να οργανώσουμε την συζήτησή μας στην πρώτη συνεδρίαση μετά το καλοκαίρι και μετά τον Σεπτέμβριο θα έχουμε τις τροπολογίες και τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων επιτροπών για να οριστικοποιήσουμε τα πράγματα. Ε, θα επισκεφτούμε και την Ιαπωνία οπωσδήποτε τον ε, Σεπτέμβριο και μετά βεβαίως ε, η ψηφοφορία προγραμματίζεται τον Οκτώβριο ή αρχές ε, Νοεμβρίου και ολομέλεια μέχρι τον Δεκέμβριο. Ωραιότατα και καλή τύχη σας εύχομαι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να τα καταφέρουμε φέτος. Ουκρανία 20 ε, Μαρτίου συγκεκριμένα συζητήθηκε η εφαρμογή της συμφωνίας ε, Ελευθερία Βορείου και η πολυμερής ε, συμφωνία και η πρώτη ε, η οποία δεν δόθηκε θα θυμάστε η τρίτη δόση γιατί δεν είχαν εκπληρωθεί κάποια όρη και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό προσεχώς γιατί υπάρχει μία νέα πρόταση της Κομισιόν Ινδονησία David Martin 21 Μαρτίου ναι ναι επί του πιεστηρίου Χτες ε, είχαμε μία ενημέρωση από την Κομισιόν ε, για την συνάντηση που έλαβε χώρα 19 με 21 Φεβρουαρίου και από την Κομισιόν αντιληφθήκαμε πως η ατμόσφαιρα ήταν ε, ικανοποιητική. Υπάρχει διάθεση για να σημειωθεί πρόοδος, αλλά η πρόοδος εξακολουθεί να είναι αργή δεν ε, είναι κάποια ανταλλαγή, κάποια συζήτηση για τους δασμούς. Ελπίζουμε να γίνει τον επόμενο μήνα και να υπάρξει κάποια πρόσφορα για τις υπηρεσίες από την άλλη. Είχαμε μια καλή πρόοδο για την ενέργεια, τις πρωτεσίλες, ε, το ειδικευμένο σύστημα προτιμήσεων. Ναι, στο θέμα του επενδυτικού δικαστηρίου το θέμα θα ληφθεί σε υψηλό επίπεδο της κυβέρνησης της Ινδονησίας. Για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη μοιάζουν δύσκολα τα πράγματα γιατί αφενός ε, είναι ανοιχτή να δεχτούν τα όσα λέμε για τις προδιαγραφές του περιβάλλοντος και τα εργασιακά και να υπάρχει μια προσέγγιση που θα βασίζεται στις κυρώσεις, αλλά, αλλά εάν και μόνο αυτό θα έχει οικονομικό όφελος. Τώρα δεν ξέρω πώς σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ούτε και ο διαπραγματευτής μας το έχει αντιληφθεί. Για τις προμηθείες επίσης είναι μόνο μία συζήτηση. Ε, το θέμα του Φινικελαίου αναφέρθηκε, δεν θα το επαναλάβω. Νομίζω καλό ήταν να γίνει μια ειδική συζήτηση για το θέμα αυτό. Από την άλλη βεβαίως ξεπλάγει που η Κομισιόν ε, είπε ότι ετέθη το ζήτημα στις συναντήσεις παρά τα όσα λοιπόν διαβάσαμε δεν υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση από την Ινδονησία όσο θα περίμενε κανείς χάρη που ο Μπας Άικχαουτ ε, ο Κόκκινος, κόκκινος εννοώ ότι ήταν υπεύθυνο για την αναδιατύπωση. Ήταν εκεί πέρα και μπορούσε να εξηγήσει την άποψη του Κοινοβουλίου. Και νομίζω πως είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διάλογοι δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι γίνεται. Συνολικά λοιπόν μια επικοδομητική συνεδρίαση, κάποια πρόοδος αλλά οι διαπραγματεύσεις κινούνται αρκετά σιγά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και στις 21 Μαρτίου υπήρχε και μία συνάντηση για την Ρωσία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει... Δεν έχουμε έντονες εμπορικές σχέσεις για διάφορους λόγους. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 21. εξέταση άμεσων ξένων επενδύσεων και να δώσω απευθεία το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Προύστ, για να μας παρουσιάσει το σχέδιο κειμένου του. Bien, merci, monsieur le, le président. Euh, Ευχαριστώ. Πριν να αρχίσω να μιλάω για την έκθεσή μου, ξέρετε ότι ήθελα να συντάξω ένα έγγραφο εργασίας προκατακτικά επειδή ε, θεωρούσα ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία ελέγχου και για να είμαστε πλήρεις, <clears throat> σας έστειλα αυτό το έγγραφο, το λάβατε και εκεί εξέτασα τα οριζόντια ζητήματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσω σε αυτό το στάδιο και τους σκιώδεις εισηγητές που εμπλούτησαν το κείμενο με, τη, με τις παρατηρήσεις τους. Προσπάθησα πραγματικά στο μέτρο του δυνατού να λάβω υπόψη τα σχόλιά τους. Ας περάσω στο σχέδιο έκθεσης ε, και στις 73 ε, τροπολογίες συγκεκριμένα που κατέθεσα. Ε, ευρωπαϊκό φιλτράσμα των επενδύσεων. Αυτό είναι το θέμα. Θα υπάρχουν πολύ μεγάλες ανταλλαγές απόψεων και για μένα υπάρχει ένα τρίπτυχο. Ε, η ε, συλλογή, η ανάλυση και ε, η διάδοση των πληροφοριών. Θα δείτε ότι σε όλες αυτές τις τροπολογίες καταθέτω προτάσεις ακριβώς για να προωθήσω αυτό το τρίπτυχο. Χωρίς όμως να θέσω ένα αμφιβόλο εξίσου σημαντικά ζητήματα. Κατά πρώτο λόγο πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στις επενδύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις διάφορες τεχνικές συγγνώμη ακροάσεις που έγιναν. Είδαμε ότι συμμετείχαν εκεί εννέα κράτη-μέλη και με τις εμπειρίες τους έδειξαν ότι όταν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός screening, ε, ελέγχου, δεν ε, ε, συνεπάγεται αυτό αυτόματα αντίκτυπο επί των επενδύσεων. Ξαναλέω, πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί σε επενδύσεις. Δεν είμαστε κατά των επενδύσεων, είμαστε κατά των περίεργων λόγω των επενδύσεων που δεν υπακούν σε κάποια οικονομική λογική, αλλά σε μια πολιτική λογική. Δεν υπάρχει ε, ε, ίχνος προστατευτισμού μέσα στις τροπολογίες. Τι σημαίνει προστατευτισμός για μένα, να προστατεύει κανείς σε αυτόν ε, για τους ε, λάθους λόγους. Όχι. Ε, εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε την τάξη και την ασφάλεια. Τα κράτη-μέλη έχουν τον τελικό λόγο για τις επενδύσεις που γίνονται στην επικράτειά τους. Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση εγώ δεν ε, θέτω να φόλο την ε, επικουρικότητα, την αρχή της επικουρικότητας, ε, η αρμόδια οντότητα που ενφύνει λαμβάνει την απόφαση είναι το κράτος. Κανέναν δεν υποχρεώνουμε επίσης να θεσπίσει μηχανισμό ελέγχου. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε ε, η συλλογή, η ποιότητα της συλλογής να χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία για να είναι και ομοιογενή τα αποτελέσματα, τα δεδομένα. Υπάρχει όμως περιθώριο λιγμών. Δεν υποχρεώνουμε κανέναν. Ε, υπενθυμίζω, 13 κράτη-μέλη σήμερα έχουν ήδη μηχανισμό ελεγκτικό. Ε, δεν υποχρεώνουμε κανέναν λοιπόν να θεσπίσει τέτοιο μηχανισμό. Ε, επιδιώκουμε ισορροπία επίσης ε, με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και να μην ε, φτιάξουμε ένα τέρας, δηλαδή θέλουμε να είναι πραγμα... ρεαλιστικός και αποτελεσματικός και σαφής ο μηχανισμός. Ε, τώρα, σχεδιαγραφώντα τις προτάσεις μου, ε, θα έλεγα ότι αρχίζοντας με το άρθρο 7, παραδοσιακή προστασία κατά των επενδύσεων ε, που δεν σχετίζονται με την πολιτική και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε, αυτό το, αυτή η γραφική αναπαράσταση σας εξηγεί πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα. Όταν υπάρχει μηχανισμός screening, κοινοποιείται στην Επιτροπή, τα κράτη έχουν 25 ε, μέρες για να ε, χνομοδοτήσουν. Ε, άλλες 25 έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συν 10 για να εκδώσει γνωμοδότηση και αποφάσισα να μειώσω κατά ένα δεκαπενθήμερο τις διορίες για να είμαστε αποτελεσματικότεροι, διότι ξέρουμε ότι σήμερα στον οικονομικό κόσμο, όπως έχει διαμορφωθεί, πρέπει να έχουμε ταχύες αντιδράσεις. Είναι το α και το ω. Αυτή η διαδικασία ε, είναι σαφής και απλή. Αυτό το πλεονέκτημα έχει. Πάμε στη σελίδα 4. Προσθέτω εδώ ένα καινούριο στοιχείο τα κράτη-μέλη που δεν έχουν μηχανισμό ή ε, που ο μηχανισμός, ο ελεγκτικός ε, δεν είναι ικανοποιητικός, δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν καλύπτονται όλοι οι τομείς από αυτόν τον μηχανισμό. Οπότε αν για μια συγκεκριμένη επένδυση ή ξένη επένδυση δεν μπορεί να ε, βγει απόφαση από αυτόν τον μηχανισμό, μπορεί σε θελού σε βάση το κράτος μέλος να ζητήσει από την Επιτροπή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος μια γνωμοδότηση. Έτσι μπορεί να ε, πάρει ε, πληροφορίες χωρίς αντίτιμο για ε, το θέμα που τον ενδιαφέρει. Για τις διορίες δεν αλλάζουμε τίποτα. Βασιζόμαστε στο προηγούμενο, στην προηγούμενη παράσταση. Πάμε τώρα στο άρθρο 9. Ποια είναι η διαδικασία όταν ε, σχετίζεται η επένδυση με πολιτική ή προγράμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς ε, ταυτόσιμη ε, λειτουργία των μηχανισμού δίνεται να εκδώσουν γνωμοδοτήσεις στα κράτη-μέλη. Γιατί, διότι χρηματοδοτούν, συμβάλλουν με κονδύλια για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνω και κάτι άλλο εγώ. Ε, να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άμεσα να ζητήσει από την Επιτροπή να εκδώσει μια χρονοδότηση και το βλέπετε ότι ζητάω ενισχυμένη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια. Σελίδα 7 τα κράτη-μέλη που δεν έχουν μηχανισμό ή όπου ο μηχανισμός δεν είναι αρμόδιος για ένα συγκεκριμένο ζήτημα μπορούν, ε, ε, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν γνωμοδότηση από την Επιτροπή ή τα άλλα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη μπορούν και αυτοβούλως να εκδώσουν την γνωμοδότηση. Οποιοδήποτε στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να εκδώσουν την γνωμοδότηση, λοιπόν, στον πυρήνα αυτή τη πρόταση λοιπόν αυτό βρίσκεται. Δηλαδή, όσο περισσότερο λιγότερες εξαιρέσεις υπάρχουν, όσο πιο ειδικές διατάξεις υπάρχουν, τόσο περιπλέκεται και ε, η γραφική παράσταση. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό εννοούσα. Πρέπει να είναι σαφής ε, και αποτελεσματικός ο μηχανισμός ε, και όχι να φτιάξουμε ένα εξάμβλωμα που αντιβαίνει στους στόχους μας. Δηλαδή να έχουμε ρεαλιστικό και αποτελεσματικό μηχανισμό που λειτουργεί ταχαίως. Το είδαμε και σε άλλες επιτροπές, στην Επιτροπή Μεταφορών. Γι' αυτό και αν το αναθεωρούν ε, μετά ε, από 10 χρόνια, γιατί είναι τόσο περίπλοκος ο μηχανισμός που ε, δεν, μπορούμε, δεν μπορούν οι χρήστε να υποφεληθούν από αυτό. Δεν μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει. Αυτό αντιβαίνει στους στόχους μας. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των επιχειρήσεων. Για τις τροπολογίες μου τι άλλο, ε, ε, ποιο άλλο σημαντικό στοιχείο υπάρχει. Σε σχέση με τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνω ένα τρίτο σενάριο. Έχουμε τα δύο σενάρια για τι νομοδοτήσεις, όπω είπαμε. Ε, βλέπετε τώρα μια γραφική αναπαράσταση τη τρίτη τρίτης ε, μου. Αν ναι ε, κάποιο επιτροπή ή κράτο μέλο θεωρεί ότι μία επένδυση συνιστά ε, απειλή για την ασφάλειά του ε, ή ε, ναι, αντιβαίνει στην πολιτική, σε μια πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη και να βρει μία λύση. Πρέπει τον λόγο κράτο μέλο, είναι σημαντική η διατύπωση, να βρει μία εναλλακτική λύση σε σχέση με την απλή έγκριση τη ξένη επένδυση. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό, είναι βεβαίω σπάνια περίπτωση αυτή, αλλά θα πρέπει να την καλύψουμε. Ε, ε αν σε περίπτωση που με μία επένδυση δημιουργεί ε, ως προς την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη πραγματικό πρόβλημα και ξέρετε ότι συμβαίνει πολύ συχνά να βλέπουμε αυτή την παθητική αντίδραση, δηλαδή διαπιστώνει κάποιος το πρόβλημα αλλά δεν κάνει τίποτα. Ε, οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την περίπτωση ολιγορίας και ε, ξαναλέω, δεν αφισβητούμε την αρχή της επικουρικότητας, γιατί η φίνε θα αποφασίσει το κράτος μέλος όπου γίνεται η ξένη επένδυση. Τι σημαίνει όμως αυτό, ότι ε, καθιδρύεται ένα σε διάλογο. Θυμάστε το τρίπτυχο στην αρχή της παρουσίαση μου, συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή. Ε, πληροφοριών. Διάλογος, ε, δηλαδή είναι ακρογωνίως λάθος, ε, συγγνώμη. είναι ε, ε, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι αυτό μπορεί να καθυσυχάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ένα κρατάς μέλος. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρει τη μορφή συνοδευτικού μέτρου, αν υπάρχει ο μηχανισμός. Εάν όχι, ε, μπορεί να σημάνει παρακολούθηση μιας απάντησης. θα δώσω ένα παράδειγμα για να <clears throat> διευκρινίσω τι σημαίνει σε αυτή την περίπτωση ξένη επένδυση σε ε, μέσω μαζικής ενημέρωσης, όπου δεν υπάρχει ε, τέτοιος μηχανισμός. Έτσι καλύπτεται η επικαιρότητα από αυτό το μέσο. Εάν ε, το κράτος μέλος επιτρέψει αυτή την επένδυση, μπορεί, ε, μάλλον μπορεί να την εγκρίνει ή ξέρω εγώ να αναθεωρήσει την ε, αδειοδότηση μετά από μια πειραματική χρονιά ή να θεσπίσει μια νομοθεσία για τις πλαστές ειδήσει. Δύο συνοδευτικά μέτρα, καταλαβαίνετε, είναι μία ε, απόπειρα να εξευρεθεί κοινή λύση, παρότι εγκρίνεται η επένδυση. Όταν έχουμε λοιπόν την ομάδα ε, παρακολούθηση των κοινών επενδύσεων και εξάλλου περιλαμβάνω όμω στον κανονισμό του, ώστε οι επιχειρήσει, τα συνδικάτα ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο ε, να εισακούεται από του εμπειρογνώμε είτε του κράτου είτε τη Επιτροπή. Για τις επόμενες προτάσεις μπορώ να πω ότι είναι ε, περίπλοκο το ζήτημα των ε, επενδύσεων και θα υπάρξουν γκρίζες ζώνες, σίγουρα. Για να καταλάβουμε υπάρχει ένα γενικό, μια γενική κορονίδα ε, που είναι η δημόσια ασφάλεια και η, η δημόσια τάξη και η ασφάλεια υπάρχουν πυλώνες τώρα και, και η γκρίζα ζώνη ανάμεσα τους ε, όπου μπορεί να εγκρίνει την επένδυση ένας κράτος γιατί θεωρείται στρατηγική αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι απαραίτητα επικίνδυνη επένδυση για την ασφάλεια για τη δημόσια τάξη. Ε, το ίδιο και για τα στοιχεία που ε, προσθέτω ως υποβοήθημα ε, για την λήψη απόφασης, αν υπάρχει αυτή η στρατηγική διάσταση της επένδυσης ή αν ξέρω εγώ, υπάρχει έλλειψη αμοιβαιότητας. Λέγαμε με την Επίτροπο ότι δεν υπάρχει αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών. Σίγουρα δεν πρόκειται για διακριτική μεταχείριση όταν χρησιμοποιούμε τέτοια κριτήρια. Ε, στα ε, πλαίσια των ανταλλαγών, του διαλόγου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το στοιχείο και είναι σημαντικό να το κάνουμε, πιστεύω εγώ για να μην υπάρχει παρανόηση. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δίνει προς τα στοιχεία προς ενημέρωση, όχι κριτήρια για να απαγορευτεί μια επένδυση. Ε, σε καμία περίπτωση και ξέρουμε αντίθετα ότι αν προτάξουμε αυτά τα κριτήρια θα αντιμετωπίσουμε ε, νομικά κολλήματα που σε σχέση με το κεκτημένο του ΠΟΕ. Ε, όμως, χάρη σε αυτέ τι πρόσθετε πληροφορίε, μπορούμε να διαμορφώσουμε μια συνολικότερη εικόνα του πλαισίου τη επένδυση. Και in fine, όπως σας έλεγα, ε, υποβοηθούνται έτσι ε, τα κράτη-μέλη να λάβουν μια απόφαση, Έχοντα όμω τα απαιτούμενα στοιχεία στη διαθέσή του για μια επένδυση που γίνεται στην επικράτεια του. Ε, ο κίνδυνο ε, παράκαμψης, η εξασφάλιση αποτελεσματικότητα, γιατί αυτό είναι ο βασικό στόχο μα. Πώ θα εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού θέλουμε αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός να επικεντρωθεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το, την πρώτη πτυχή, συλλογή πληροφοριών ε, για την, ε, ε, την ταυτοποίηση του τελικού επενδυτή, διότι συχνά τι συμβαίνει. Υπάρχει πίσω από τον ε, μια βιτρίνα πίσω από έναν επενδυτή κρύβεται ένας ολόκληρος όμιλος ε, και ε, κρύβεται η πραγματική ταυτότητα του επενδυτή. Λοιπόν, συλλογή πληροφοριών για λόγους διαφάνειας και ασφαλής να ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από τον επενδυτή, να ξέρουμε να τον ταυτοποιήσουμε. Πολύ σημαντικό αυτό το, αυτή η πτυχή, αυτή η διάσταση συλλογής πληροφοριών. Για τις στρατηγικές πληροφορίες θα το δείτε. Ε, υπάρχει διεύθυνση για να καλυφθούν όλοι οι τομεί αν υπάρχει θέμα δημόσια τάξη ασφάλεια. Ε, μετέβαινε στην ε, Ουάσιγκτον για να δω τι κάνουν οι συναδέλφοι μα ε, για τα θέματα τη ασφάλεια. Εκείνη στην νομοθεσία του τα, τα βάζουν όλα μέσα ό,τι σχετίζεται με την ασφάλεια. Όμω, εγώ πιστεύω είναι σημαντικό να παριθμίσουμε σωστά του τομεί που ενδεχομένω μπορούν να επηρεάσουν την τάξη και την ασφάλεια. Αεροναυπηγική, ε, μαζικά δεδομένα, ε, τεχνητή ε, νοημοσύνη, γεωργικέ εκμεταλλεύσει που δημιουργούν προβλήματα, ΜΜΕ ή ξέρω εγώ μπαταρίε. Ξέρετε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ε, για την στρατηγική μας, για την αυτοκινητοβιομηχανία θα μας πούνε εκείνοι. Ε, τελειώνω, τελειώνω. Ε, δημόσια έκθεση. Ε, μπορεί να είναι απλό το σύστημα και παρόλα αυτά πολύ αποτελεσματικό. Θα το αποδείξω. Θα υποβάλει έκθεση ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα, φυσικά υπάρχουν θέματα εμπιστευτικότητα και θα, θα ε, σεβαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δημοσιοποιήσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Κλείνοντας και συνοψίζοντας τις προτάσεις ε, που κάνω, που μοναδικό στόχο έχουν, ε, όπως έλεγε ο, ο διάσημος συγγραφέας Προύστ, ε, ε αναζητώντας το χαμένο χρόνο, Ε, ξέρετε ότι είμαστε η μόνη, η μόνη ε, οικονομική δύναμη στον κόσμο που δεν έχει τέτοιο ελεγκτικό μηχανισμό. Για να είναι ε, ξεκάθαρο και ρεαλιστικό ο μηχανισμό, λοιπόν, ε, ε αυτό που χρειάζεται αυτόν τον ξεκάθαρο και ρεαλιστικό μηχανισμό είναι η Ευρώπη. Και από κοινού και το τονίζω, το υπογραμμίζω αυτό, όλοι μαζί, με την Επιτροπή, με το Συμβούλιο, με τα κράτη-μέλη, οφείλουμε να βρούμε μία ε, ισόρροπη λύση ρεαλιστική και κυρίως αποτελεσματική. Σίγουρα είναι στενό το χρονοδιάγραμμα, διότι έχουμε τις εκλογές που επίκυνται και ο στόχος φυσικά είναι να βρούμε λύση μέχρι το τέλος του Πιστεύω όμως ότι αν ε, συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας και έχουμε αυτόν τον κοινό στόχο, όχι να είμαστε κατά των επενδύσεων, αλλά να είμαστε κατά των ε, περίεργων επενδύσεων, πιστεύω, είμαι πεπισμένος ότι θα βρούμε μια λύση που και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κρατών αλλά και στις ανάγκες των επιχειρήσεων γιατί πίσω από τον ελεκτικό μηχανισμό Ξέρετε, συχνά απειλούνται κλάδοι ολόκληροι. Και όταν απειλούνται κλάδοι, απειλείται ε, η απασχόληση και ξέρουμε ότι η απασχόληση για μα είναι ύψιστη προτεραιότητα. Ευχαριστώ και παραμένω στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Προύστ. Έχουμε ένα τέταρτο μόνο. Μόνο ένα τέταρτο. Και έχουμε τους κοιόδης συζητητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να ολοκληρώσει και να συνοψίσει. 1,5 λεπτό το πολύ λοιπόν. Η Μακουλάδα πρώτα για του ελθέ και δημοκράτε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί πραγματικά έκανε εξαιρετική δουλειά και εξαιρετική παρουσίαση και ελπίζω να μπορέσει να τη δώσει και σε όλα τα μέλη. Εγώ θα ήθελα να τονίσω δύο θέματα τα οποία μου φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Να βρούμε τον τελικό επενδυτή, αλλά με ποια μέσα, ε, ποιος θα τον βρει. Και δεύτερον, έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε λίγο τον αντίκτυπο ε, της απουσίας κατάλληλης νομοθεσίας, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο γίνεται αυτή η νομοθεσία, την οποία εγώ υπερασπίζομαι ε, και νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι γίνονται πάρα πολλά βήματα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, το οποίο θα σας παρουσιάσω αλλά ε, πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να υπά... λογικά να υπάρξουν και αντιστάσεις από κάποια κράτη-μέλη και θα πρέπει να έχουμε μια καλή μελέτη αντικτύπου ε, να τη δώσει, να τις δει στο κοινοβούλιο, γιατί νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλη δουλειά να κάνουμε, μακρά πορεία. Και κάτι ακόμα, και με αυτό ολοκληρώνω. Μπορούμε να συσχετίσουμε τη διαδραγμάτευση συμφωνών επενδύσεων με τρίτες χώρες ε, με μια δέσμευση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Σταρμπάτη. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή. Θα θέλαμε και την παρουσίασή σας, η οποία ήταν πολύ αναλυτική. Γι' αυτό μπορώ να είμαι σύντομος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πραγματική την κατάσταση στην ε, κάθε χώρα, κάποιες είναι πιο περιοριστικές, κάποιες πιο ανοιχτές, έχουμε την ιστορική εμπειρία, αλλά μας διαβεβαιώσατε πως θα ισχύει η αρχή της επικουρικότητας και είναι σαφές κάθε χώρα ξέρει καλύτερα το τι είναι ευνοϊκό οπότε ας δούμε την αξιολόγηση αντικτύπου πάντα βεβαίως ε, οι επενδύσεις από το εξωτερικό είναι καλές όταν πληρούν κάποιους όρους ε, και οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι εντό του πλαισίου του ΠΟΕ να μην ε, περιέχουν αυτά τα οποία αναφέρεται ως αρνητικά στοιχεία. Ακριβώ θα πρέπει να δούμε το τι θα κάνουμε και εμείς... Ε, το για πολιτικοποίηση υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, ε, θα πρέπει λοιπόν να τον αποφύγουμε. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια μορφή διεθνούς κατανομής εργασίας. Μια ερώτηση ακόμα. Ε, τεθεί το ζήτημα της αμοιβαιότητας ε, σε σχέση με κάποιες χώρες οι οποίες εκμεταλλεύονται τα πράγματα ξετσίποτα. Και ε, το θέμα είναι μετά τι ζητάνε από μας. Οπότε θα έπρεπε ακριβώς να δούμε ίσως το τι μπορεί να γίνει με αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην αμοιβαιότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Χαράντσοβα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εκθεσή του. Έχω αρκετά σχόλια, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πέντε πράγματα θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοιχτεί όσο ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις όσο είναι σήμερα. Οι επενδύσεις είναι μία από τις βασικές ε, δυνατότητε, δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ κατά τον καθορισμό αυτής της νομοθεσία και να λάβουμε δεόντως υπόψη τη νομική του βάση. Αυτό ο κανονισμό πλαίσιο βασίζεται στη δημόσια ασφάλεια και στη δημόσια τάξη και επομένω δεν θα πρέπει να είναι εργαλείο για να κλείσουμε τις αγορές μας ε, ε, για λόγου αμοιβαιότητα οικονομικών συμφερόντων. Τρίτον, όπως παρουσιάστηκε η πρόταση δεν είναι μόνο επιπλέον διοικητικό άχθος για τις διοικήσεις των κρατών μελών αλλά θα μπορούσε να έχει και παρέμβαση των κρατών μελών ε, στις διαδικασίες ε, της κάθε χώρας. Ε, πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να ε, ελέγχουν ε, στη διακριτική τους ευχαίρεια, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε υποχρεώσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέραν των όσων περιλαμβάνονται στην αρχική της πρόταση. Τέταρτον, χαίρομαι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και να συσταθεί και μια σχετική ομάδα συντονισμού. Πιστεύω ότι η έκθεση θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τα θέματα αυτά. Σίγουρα υπάρχει λόγο συντονισμού, αλλά ταυτόχρονα η εξουσία λήψης αποφάσεων θα πρέπει να είναι στα κράτη-μέλη και στι αρμόδιε αρχέ. Τέλος, για τους διάφορου τομεί. συνειδητοποιώ ότι ο εισηγητή διεύρυνε κατά πολύ του τομεί αυτή. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι τέτοιο και νομίζω ότι κάποιοι από τους τομεί ε, δεν είναι ε, κατάλληλοι και δεν πρέπει να αναφέρονται, αλλά υπάρχει ένα που θα ήθελα να αναφέρω, το μέσο μέσων ενημέρωση. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι ο ρόλος είναι κομβικός και στρατηγική σημασία για την κοινωνία και για τις ε, δημοκρατικές διαδικασίες, επομένως θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Ευχαριστώ. Η Τιτσιάνα Μπεγκίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά του. χρειάζεται να γίνεται έλεγχο ε, των διεθνών επενδύσεων για να μην υπάρχει υπερβολική συσσόρευση εξουσία και να μην ε, ε, επιτρέπουμε σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν δρούν πάντα προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να συγκεντρώνουν πολλές δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και για την υδροδότηση κλπ. Δεν μας ικανοποιεί όμως ο τομέας της άμυνας, διότι όταν δεν υπάρχει εθνικός έλεγχος των ξένων επενδύσεων, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητήσουμε από όλε τι χώρε μέλη που δεν έχουν να έχουν ένα σύστημα εθνικού ελέγχου των ξένων επενδύσεων Σίγουρα συμφωνούμε ότι ένα από τα κριτήρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη για τα ε, ξένες επενδύσεις είναι το κριτήριο της αμοιβαιότητα και η πρότασή μας είναι να προβλέψουμε και παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να ελέγξουμε ποιος είναι ο, ο τελικός ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης που κάνει μια επένδυση και να επαληθέσουμε αν πρόκειται για ένα πραγματικό οικονομικό φορέα ή για κάποια ξένη ε, κυβέρνηση η για καποια ξενη προσπαθεί να επιτύχει τις πολιτικές της επιδιώξει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ότι πρέπει να εξετάζεται μια επένδυση όχι μόνο από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τους πολίτες, από την κοινωνία των πολιτών και από τους ενδιαφερομένους. Έχουμε διάθεση συνεργασίας και φυσικά ε, θα προτείνουμε και θα ε, καταθέσουμε και τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούχνερ. Ε, δεν είμαι εγώ σκιώδης εισηγητής. Είμαι όμως ο μιας επιτροπής που γνωμοδοτεί. Τα σημαντικά ακούστηκαν. Θα ήθελα όμως να προσθέσω το τι μας ενδιαφέρει από την σκοπιά της ΣΕΝΤΕΤ. Έχουμε το θέμα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και των τεχνολογιών κλειδί θα ήθελα εδώ πέρα να επιθυμίσω την περίπτωση της εταιρείας Κούκα στο Augsburg που αγοράστηκε η εταιρεία από μια κινέζικη εταιρεία η οποία εταιρεία Κούκα ήταν πρώτη στον κόσμο στην τεχνολογία της η οποία μεταβιβάστηκε στην Κίνα και τελικά εισάγουμε την τεχνολογία αυτή εμείς από την Κίνα. Πρέπει να αποφευχθούν αυτά στο μέλλον είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να ανταλλάξουμε πληροφορίες ε, για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ε, το χρειαζόμαστε αυτό για να γνωρίζουμε το τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τις επενδύσεις ε, τις οποίες δεν θέλουμε. Και ο Πέντρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα σύντομο σχόλιο. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ τον εισηγητή Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν είναι λογικό αυτό το χρονοδιάγραμμα δεδομένων των όσων ε, έχουμε μπροστά μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν ε, χρειάζεται αυτό το τόσο σύντομο χρονοδιάγραμμα για τις ε, τροπολογίες. Η Κομισιόν πέντε λεπτά το πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Περίμενα να μου δώσετε λιγότερο χρόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι και πιο γρήγορη. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και για τον επαγγελματισμό του επαγγελματισμό αυτής της ανάλυσης ε, φαντάζομαι δεν θα σας προξενήσει η έκπληξη το να πούμε ότι το θέμα αυτό είναι θέμα προτεραιότητα για την Κομισιόν και είναι ένα θέμα στο οποίο θέλουμε να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο πριν από το τέλος της θητείας αυτής. Ταυτόχρονα έχουμε μπροστά μας δύσκολη δουλειά και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τρόπο ρεαλιστικό και γρήγορο. Ε, δεν έχουν προχωρήσει ακόμα τα πράγματα. Πρέπει να συνεργαστούμε και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και το σημαντικό είναι να μην ε, ξεχάσουμε εδώ πέρα τον βασικό στόχο αυτής της πρότασης Πρέπει δηλαδή να είμαστε εξοπλισμένοι με μέσα τα οποία θα μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Να δούμε τις συναλλαγές ε, που γίνονται στις ε, αγορές μας ε, για επενδύσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στην Ευρώπη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επενδύσουμε την ασφάλεια όχι μόνο των κρατών μελών αλλά ολόκληρης της Ένωσης. Αυτό είναι μια νέα προσέγγιση και το αναγνωρίζω αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης σημαντικό είναι να έχουμε κατά νου ότι είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα. Είναι κάτι καινούργιο. θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα εάν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη δεσμεύονται όχι μόνο στην ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και μεταξύ τους και με την Κομισιόν κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και βεβαίως ε, πρέπει να έχουμε κατά νου ακριβώς ε, το ότι υπάρχουν και άλλες χώρες στον ε, κόσμο που έχουν τέτοια συστήματα και εξετάζουν αν υπάρχει ανάγκη να τα ενημερώσουν και βεβαίως να σκεφτούμε την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας όπως ακριβώς τώρα ε, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ανάγκη να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη, πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλες χώρες στον κόσμο. Αυτό είναι κάτι ε, όπου πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει και για αυτόν τον σκοπό χρειάζεται αυτός ο κανονισμός. Πολλά πράγματα έχουν ακουστεί στις διάφορες παρεμβάσεις, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, αλλά θα ήθελα να επιμείνω σε δύο βασικά αλλά πολύ σημαντικά πράγματα, δύο αρχές που πρέπει να μας καθοδηγούν εδώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο έλεγχος ε, των άμεσων ξένων επενδύσεων δεν θα γίνει ένα μέσο ε, προστατευτισμού δεν θα ανοίξουμε έτσι πόρτες για τους Ευρωπαίους επενδυτές αλλού και πρέπει να είναι ανοιχτέ οι πόρτες για τους Ευρωπαίους επενδυτές. Επίσης αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθήσαμε και στους μηχανισμούς που υπάρχουν ήδη στα κράτη-μέλη μας. Αυτά λοιπόν λειτουργούν ε, με βάση την ασφάλεια και την δημόσια τάξη και πρέπει να αναφέρουμε ότι ο τελευταίος λόγος βεβαίως πάντα ανήκει στα κράτη-μέλη. Ε, αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Είμαστε διαφορετικά κράτη-μέλη με διαφορετικές ανησυχίες. Σταματάω λοιπόν εδώ. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή και σας ε, για την γενναιοδορία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρόνο γιατί έχουμε και περιορισμό, πρέπει να τελειώσουμε στη μία Κύριε Σιγητά, υπήρχε ένα αίτημα να δοθεί λίγο περισσότερη διορία για τις τροπολογίες. Μπορούμε να έχουμε τροπολογίες ε, στις 4 Απριλίου, αλλά μετά δεν έχουμε εγγύηση ότι θα μεταφραστούν όλες οι ε, τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες. Οι βασικές γλώσσες βέβαια συζήτησης θα μεταφραστούν, αλλά ε, για την επόμενη συνεδρίαση και ψηφοφορία θα γίνει στις 17 Μαΐου. Ε, μπορεί να κάνετε λοιπόν ένα δωράκι στους συναδέλφους και να τους δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο. Τι γνώμη έχετε. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, δεν έχω πρόβλημα να προσθέσουμε μερικές μέρες στην προθεσμία αλλά είναι αλήθεια ότι ξεκινά μια περίοδος με αρκετές μέρες αργίας και αν θέλουμε να τηρήσουμε την ε, ημερομηνία ψηφοφορίας θα πρέπει πραγματικά να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε λίγο καλύτερα στην ανησυχία σας όσον αφορά τις προθεσμίες γιατί για άλλη μια φορά όπως σας είπα στην εισαγωγή είναι ένα περίπλοκο θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε και αν θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποιο καλό συμβιβασμό ε, να δώσουμε ένα επιπλέον χρόνο λαμβάνοντας υπόψη και τις μέρες της αργίας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε καιρούς στις 17 Μαΐου. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ήδη ασχολούμαστε λίγο με το κείμενο και να ευχαριστήσω κυρίως ε, και για την ε, διάθεση και την ε, όρεξη που έδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει διάλογος και μια πραγματική λύση διότι για άλλη μια φορά είναι πράγματι ότι όταν μας ακούνε, έφυγε βέβαια συνάδελφος για την αμεβαιότητα ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει τουλάχιστον ε, να ξαναδούμε καλά αυτή την έκθεση και δεν ξέρω αν ο όρος αμοιβαιότητα ε, μπορεί να περιληφθεί στα κριτήρια διάκρισης, διότι είχαμε μια τεχνική ακρόαση με την Ιταλία και είχαν συμπεριλάβει την αμοιβαιότητα στη δική τους τη διαδικασία screening και ε, τους επανέφεραν στην τάξη διότι δεν ήταν σωστή αυτή η προσθήκη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι επειδή για άλλη μια φορά αυτή η έκθεση βασίζεται στο διάλογο και στην ανταλλαγή ε, απόψεων, τίποτα δεν απαγορεύει στα κράτη-μέλη ή την Κομισιόν να πούνε ότι υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας, δυσκολία αμοιβαιότητας στα πλαίσια διαλόγου και σε γενικές γραμμές ε, να μπορέσουμε να τα έχουμε αυτά για μια χώρα, αλλά δεν μπορούμε να το συμπεριλάβουμε και δεν μπορεί να εμφανίζεται ως ένα κριτήριο ξεχωριστό, διότι δεν θα συνάδει αυτό με τους κανόνες. Για την Ισπανίδα συνάδελφο. Πράγματι, η μελέτη δικτύπου είναι ένα θέμα το οποίο ετέθη. Θα απαντήσουμε αργότερα. Εντάξει, θα τα πούμε διμερώς. Ευχαριστώ για την ε, συμβολή σα και ε, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Προύστ. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 4 Απριλίου, 6 ώρα. 4 Απριλίου, 6 ώρα. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες στην επόμενη συνεδρίαση. 23 και 24 Απριλίου και ψηφοφορία 17 Μαΐου. Σημείο 22, τίποτα στα διάφορα. 23, επόμενη συνεδρίαση, 23 και 24 Απριλίου. Καλό Πάσχα.